επίτροπος απαντήσει βάσει αρχής ping-pong, δηλαδη δηλαδή ε, ερώτηση-απάντηση και ούτω καθεξής. Θα ξεκινήσουμε με ένα γύρο ερωτήσεων από τους επικεφαλείς των 7 πολιτικών ομάδων προς την Επίτροπο. Και ο καθένας θα έχει 7 λεπτά, 1 λεπτό για ερώτηση, 2 λεπτά απάντηση, 2 λεπτά συμπληρωματική ερώτηση, ένα λεπτό απάντηση. Στο δεύτερο γύρο θα υπάρξουν 38 ερωτήσεις με ε, τρία λεπτά ε, κάθε μία, δύο λεπτά για την ερώτηση και ένα λεπτό για την απάντηση. Στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στον κύριο Λεμπρούν, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Περιφερειών, για μια σύντομη δήλωση. Στο τέλος, η κυρία Κορίνα Κρέτσου, υποψηφία επίτροπος για την περιφερειακή πολιτική, θα έχει πέντε λεπτά, χρονοφυρίδα πέντε λεπτών για τις ε, καταληκτικές της παρατηρήσεις. Ο καταμερισμός του χρόνου αγόρευσης ακολουθεί τη μέθοδο DONT, βάσει το οποίο η, τάξη, η σειρά των παρεμβάσεων έχει αποφασιστεί από τις πολιτικές ομάδες. Οι ερωτήσεις δεν, είναι, ε, δεν κατηγοριοποιούνται αναθέματα. Ε, θα πρέπει να τονίσω ότι είναι ουσιαστικό όλοι οι ομιλητές να τηρήσουν τα χρονικά όρια για τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις, γιατί αν όχι δεν θα έχουμε, θα ξεπεράσουμε το χρόνο μας και ορισμένα μέλη δεν θα έχουν δυνατότητα να πάρουν το λόγο. Ακριβώς όπως στην Ολομέλεια, ένα ρολόι θα, θα δείχνει πόση ώρα έχετε μιλήσει. Έχουμε διερμηνία στις 23 γλώσσες. Όλοι οι ομιλητές μπορούν λοιπόν να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα τους, αλλά παρακαλώ να μην μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα. Και τώρα μετά από αυτές τις παρατηρήσεις Ελπίζω ότι η διαδικασία είναι ξεκάθαρη για όλους και ε, θα κηρύξω την έναρξη της συνεδρίασης και θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στην υποψηφία επίτροπο για μια παρουσίαση η οποία δεν θα ξεπεράσει τα 15 λεπτά. Αυτή η παρουσίαση θα ακολουθεί από χρόνο υποβολής ερωτήσεων και απαντήσεων εκ μέρους της κυρίας Κρέτσου. Παρακαλώ κυρία Κρέτσου. Ε, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι υποψήφια επίτροπος για την περιφερειακή ε, πολιτική και θέλω να ζητήσω την υποστήριξή σας. Ξέρω την διαδικασία διαπραγμάτευσης για το νέο νομοθετικό πλαίσιο και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές γιατί ε, καταβάλατε μια συλλογική προσπάθεια μετά από μια διετή διαδικασία διαπραγματεύσεων έχουμε ένα νομοθετικό ε, πακέτο. Επίσης υπάρχουν ε, νέα μέλη που έχουν μεγάλη επιτόπια πείρα και θα δώσουν προστιθέμενη αξία στην εργασία μας τα επόμενα έτη. Επίσης θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμή στον Επίτροπο Χαν, ο οποίος πραγματικά αναθεώρησε και μεταρρύθμισε αυτή την πολιτική. Η περιφερειακή πολιτική δείχνει την αλληλεγγύη μας μέσα στα πλαίσια του προτύπου κοινωνικής αγοράς και επειδή σήμερα αποζητούμε να βγούμε από την κρίση, η περιφερειακή πολιτική θα υποστηρίξει τις επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Μας δίνει την ε, δυνατότητα να αποστείλουμε ένα μήνυμα ως προς τα ευεργετήματα της ολοκλήρωσης στο Βορρά και Νότο, στην Ανατολή και τη Δύση, τη στιγμή που ολοκληρώνουμε την ανταγωνιστική οικονομία για όλους τους πολίτες. Γι' αυτό πιστεύω ότι η περιφερειακή πολιτική θα συνεισφέρει στην ε, εργασία του κυρίου Γιούνκερ ως προς την, ε, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη μέσα στα πλαίσια της ε, πολιτικής μοχλεύσεων και της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. Αυτή η πολιτική θα ορίσει και τις βασικές προτεραιότητες στον τομέα της καινοτομίας, ΜΜΕ, ψηφιακή ενιαία αγορά ενεργειακή ολοκλήρωση, κλιματικές αλλαγές, διευρωπαϊκά δίκτυα και ε, εξάλληψη του κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης, λαμβάνει υπόψη τις ε, περιφερειακές ε, και τοπικές συνθήκες και αρχές σε σχέση με το τι επικρατεί είτε στις πρωτεύουσες είτε στις πιο απομακρυσμένες περιοχές θα συμπεριλάβουμε και τους τοπικούς παράγοντες καθώς και τους περιφερειακούς. Μιλάμε για 270 περιφέρειες και 500, 500 εκατομμύρια πολίτες, πάνω από 500 εκατομμύρια. Χρειάζεται υποστήριξη του προϋπολογισμού. Δεν πρόκειται για φιλανθρωπία από τους πλούσιους στους φτωχούς. Είμαι πεπισμένη ότι επενδύοντας την πραγματική οικονομία στους ανθρώπους, στις περιφέρειες, εάν τους βοηθήσουμε, τότε η ευρωπαϊκή οικονομία θα καταστεί πιο εύρωστη και φυσικά το σύνολο είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των μερών του. Ως προς τις ε, πολιτικές μου προτεραιότητες, αν διοριστώ. Καταρχήν, θα ήθελα να εξασφαλίσω, να βελτιστοποιήσουμε την ε, ε, συμμετοχή της περιφερειακής πολιτικής για δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης. Επίσης, η μεταρρύθμιση όρισε τον επενδυτικό πυλώνα της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Επίσης θέλουμε να φτάσουμε σε αποτελέσματα για να βγούμε από την κρίση. Θα πρέπει να διαπραγματευτούμε ε, λειτουργικά προγράμματα, επιχειρησιακά προγράμματα τα επόμενα 7 χρόνια και θα πρέπει ε, να ε, προωθήσουμε τις ΣΟΕΣ οι οποίες θα δώσουν θα κάνουν τη διαφορά για την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών, για τους άνεργους και για τα εδάφη και τις περιφέρειες που μπορούν πιο εύκολα να αποδομηθούν. Θα ήθελα να πω ότι η ποιοτική, ο ποιοτικός προγραμματισμός δεν θα πρέπει να διακυβευτεί. Άρα το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική πολιτική, μεγαλύτερη αποδοτικότητα, έτσι ώστε οι νέες αρχές ερεσιμότητας να τηρηθούν με βάση τις ε, ευρωπαϊκές ε, προπτικές και το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης. Τη στιγμή που οι δημόσιοι πόροι, οι εξασθενούν, τα καλύτερα προγράμματα σημαίνουν μεγαλύτερη απασχόληση και ανάπτυξη. Αυτό θα ήθελα να το κάνω σε στενή συνεργασία με τους υπεύθυνου ε, συναδέλφους για την τομεακή αυτή ε, πολιτική, επιζητώντας συνέργειες και υποστήριξη από κοινοτικές ε, δράσεις. Θα ήθελα να με υποστηρίξετε Επίσης, αποστέλλοντας ένα μήνυμα στα κράτη-μέλη, η περίοδος προγραμματισμού 14-20 δεν αφορά ένα πρότυπο business as usual. Έχουμε μία μοναδική ευκαιρία και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και το τελευταίο ευρώ του προϋπολογισμού. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και όσον αφορά τις υποχρεώσεις νομίζω ότι οι βασικοί δικαιούχοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο τα χρήματα που λαμβάνουν. Πρόκειται για τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Θα πρέπει να δείξουμε τη δέσμευσή μας στο ευρωπαϊκό, στον ευρωπαϊκό προγραμματισμό με αυτά αποτελέσματα. Μαζί είμαστε πολύ πιο δυνατοί. Όπως προβλέπετε από τον κανονισμό θα υποβάλλω στην Ρέτζη του χρόνου την έκθεση της έκβασης των διαπραγματεύσεων, αν διοριστώ. Ως προς την βέλτιστη διακυβέρνηση και την ε, θεσμική δυναμική και ικανότητα, πιστεύω ότι το θέμα είναι πολύ πιο σημαντικό από τα χρήματα και απαράβατος όρος για να επιτύχουμε. Θα πρέπει να έχουμε πολύ καλή διοίκηση διοικητικά μέσα, ιδιαίτερα στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει υποστήριξη για τη θεσμική ικανότητα στα νέα, με τα νέα προγράμματα και να υποστηρίξουμε τα κράτη κατά την επόμενη περίοδο. Χρειάζονται εταιρικές σχέσεις και συνέργεια δημόσιου ιδιωτικού τομέα Επίσης χρειάζονται εταιρικέ σχέσεις υψηλής ποιότητας για τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων. Πολλά μπορούμε να μάθουμε από τις βέλτιστες πρακτικές των περιφερειών, των πόλεων, των τοπικών αρχών και των ΜΚΙο. Θα κάνω πλήρη χρήση των νέων δυνατοτήτων από το, τα αστικά δίκτυα μέσα στα πλαίσια της ανταλλαγής ε, εμπειριών. Επίσης, δεν απλουστεύουμε πάντα τις πολιτικές μας υπέρ των δικαιούχων και γι' αυτό θα πρέπει να ε, εισακουστούν οι ΜΜΕ μέσω της υποστήριξης με αυτή την ε, πολιτική, γιατί πολλές φορές υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία. Το ρυθμιστικό πλαίσιο δίνει δυνατότητες να υποστηρίξουμε τους δικαιούχους και θα συνεργαστώ με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να τηρηθούν αυτές οι αρχές. Επειδή η πολιτική συνοχή αποτελεί το 1 τρίτο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, θα προσδώσω μεγάλη σημασία στα μέτρα έτσι ώστε να υπάρχει καλή διαχείριση των διαρθρωτικών ε, ταμείων με βάση την ε, χρηστή οικονομική διαχείριση θα υπάρχει μηδενική ανοχή στην απάτη. Γι' αυτό θα ήθελα να δούμε καλύτερα την αποδοτικότητα και τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής. Θα ήθελα να συνεργαστώ με την Επιτροπή σας για να δω πώς μπορούμε να δούμε αυτά τα ζητήματα σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία και με τους πολίτες, διότι νομίζω ότι δεν μπορούμε πάντα να δούμε τι ακριβώς ε, κάνουμε. Ως προς την αποδοτικότητα της πολιτικής ε, θα ληφθεί υπόψη στο επόμενο ε, νομοθετικό πλαίσιο μετά το 2020 θα ήθελα να ξεκινήσουμε μια συζήτηση με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήδη από τα πρωταρχικά στάδια, όπως είπε και ο πρόεδρος Γιούνκερ στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές. Η ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετούς θα πρέπει να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, α, ε, ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Άρα θα ήθελα να επιδοθούμε σε έναν επικοδομητικό πολιτικό διάλογο με βάση τα, το χαρτοφυλάκιό μου για την χρηστή διακυβέρνηση. Η σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπής και Κοινοβουλίου θα πρέπει να βασίζεται στη διαφάνεια, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, σεβασμό και κοινού στόχους για να συνεργαστούμε προς συμφέρον των πολιτών. Γι' αυτό θα συνεργαστώ με σας, έτσι ώστε να φτάσουμε στους κοινού στόχους. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για μια κοινή συζήτηση και μια κοινή προσπάθεια να είναι αποτελεσματική η πολιτική αυτή. Thank you. Η Πρόεδρος Μιχαήλοβα, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κρέτσου. Ας αρχίσουμε τώρα τον πρώτο γύρο των ερωτήσεων με τον κύριο Βαν Νίστερ Ευχαριστώ πολύ κυρία Κρέτσου. Σας καλωσορίζω εξ ονόματος των μελών του Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή μας στον κόσμο της συνοχής και της περιφερικής ανάπτυξης. Νέος κόσμος για σας. Μόλις ψηφίσαμε νέους κανονισμούς με 350 δισεκατομμύρια επενδύσεις που είπατε και εσείς προηγουμένως. Έχει καλώς. Τα άσχημα νέα όμως είναι ότι η διαφορά, η απόσταση μεταξύ υποχρεώσεων και πληρωμών μεγαλώνει διαρκώς το χάσμα αυτό και οδηγεί σε προβλήματα ρευστότητας για προγράμματα που έχουν ήδη υλοποιηθεί και για τους απολύπτες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το έλλειμμα πέρσι ήταν 23,4 δισεκατομμύρια στη συνοχή και μεγαλώνει ακόμη η υποψηφία επίτροπος και η Επιτροπή γενικά. Πώς θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα αυτό. αυτοί που επωφελούνται από τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δηλαδή θα σεβαστεί τις υποχρώσεις που έχει αναλάβει. Η υποψηφία Επιτρόπος. Σας συγχαίρω για τα όσα έχετε πράξει ως μέλος της Επιτροπής, όπου είσαστε βεβαίως για τόσο μεγάλο διάστημα και έχετε συμβάλει σημαντικά στις εργασίες της. Έχετε δίκιο ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση αυτή. Μας ανησυχεί πολύ, διότι όπως είπατε τα προβλήματα για τους ε, απολύπτες της βοήθειας είναι πολύ σημαντικά και το έλλειμμα είναι πολύ μεγάλο και θα αυξηθεί μέχρι τέλους του έτους εφόσον τελικώς ε, γίνει οριστική η εκλογή μου, θα συνεργαστώ και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο Υπουργών, αλλά σας βεβαιώνω ότι θα θέσω το θέμα ενώπιον του συλλογικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι θεωρώ ότι χρειαζόμαστε όχι μόνο καλής ποιότητας προγράμματα, αλλά και σοβαρή δέσμευση χρηματοδότησης των επενδύσεων αυτών. Θα συζητήσω λοιπόν με την Επίτροπο Αρμόδια για τον προϋπολογισμό, με τους αντιπροέδρους που είναι αρμόδιοι για το πρόβλημα αυτό. Πάντως, ίσως μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς αν στηρίξετε την πρόταση διορθωτικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2015 και για το 2016. Ε, είναι σημαντικό να ανακοπεί η κατηφορική αυτή πορεία που είναι σαν χιονοστιβάδα με τους ε, απλήρωτους λογαριασμούς και πρέπει να βρούμε μια λύση, κάποια λύση για να αποφύγουμε τις συστηματικές καθυστερήσεις των ε, πληρωμών για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Όμως όπως είπα το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι ότι θα πω στους συναδέλφους μου ότι δεν είναι δυνατόν να διακινδυνεύσουν όλες οι επενδύσεις καινοτομίας, ενέργειας, για να μην μιλήσω καν για την εκπαίδευση, για τον αγώνα κατά της στόχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Είναι σημαντικό να υπάρξει η δυνατότητα να πληρωθούν οι λογαριασμοί που μένουν ακόμη απλήρωτοι. Ο κ. Βανίστερο, ευχαριστώ. Χαίρομαι που βλέπω ότι κατανοείτε το βαρύ αυτό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσετε ε, τα επόμενα χρόνια και μιλήσατε κι εσείς για αυτό το εφέ της χιονοστιβάδας. Θα πρέπει να ενημερώσετε την παρούσα Επιτροπή σε τακτική βάση. Εμείς θέλουμε να υπάρχει μια προσαρμογή, διότι είχαμε αυτή τη ροή πληροφοριών από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειών, αλλά πολύ λίγα μας λέγανε πολύ αργά, με μεγάλη καθυστέρηση και χωρίς πραγματική συζήτηση. Με τον τρόπο αυτό δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε κι εμείς στο έργο σας ούτε και να εκπληρώσουμε τα δικά μας καθήκοντα. Θα μπορέσετε λοιπόν να είστε κρυσταλλίνης διαβίας ότι θα μας δίνετε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες στην Επιτροπή μας. Μπορείτε να λάβετε δέσμευση ότι θα προσέρχεστε ενώπιον της Επιτροπής μας για να συζητείτε τα θέματα αυτά, για να γίνουν πραγματικές αλλαγές. Δεν συζητεί μονάχα η Επιτροπή Προϋπολογισμών το τι γίνεται εδώ οι ψηφοφόροι ρωτούν και σας ρωτούν και μας τι γίνεται. Μπορείτε λοιπόν να δώσετε αυτή την υπόσχεση. Από την άλλη μεριά βέβαια τη αιθούσης έλεγα τα ίδια πράγματα που λέω τώρα. Δεν πρόκειται να αλλάξω διότι και εγώ ήμουν ευρωβουλευτής. Είναι κρίσιμο λοιπόν να υπάρξει αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών και να βρεθεί λύση από κοινού. Διότι όπως είπα δεν αφορά το πρόβλημα μοναχά της περιφέρειας, αφορά ολόκληρο τον προϋπολογισμό. Προκαλεί πολλά προβλήματα επιτόπου. Και για να είμαι και ειλικρινής, δεν κατανοώ πώς είναι δυνατόν να ζητούμε από τις χώρες μέλη να πληρώνουν μέσα σε προθεσμίες ή 60-90 ημερών και εμείς να μην πληρώνουμε όλες τις υποχρεώσεις μας. Είναι σημαντικό αυτό. Θα το θέσω λοιπόν όπως είπα ενώπιον του συνόλου του Συλλογικού Σώματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γκοτσολίνο. Ευχαριστώ. Καταρχήν να σας ε, καλωσορίσω και σας εύχομαι να ανταποκριθείτε σε αυτή την εργασία. Εξ των σοσιαλιστών ε, και δημοκρατών ξέρουμε τη δραστηριότητά σας ως ε, ευρωβουλευτή. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα πρόβλημα που ανακύπτει από τις πρώτες εταιρικέ σχέσεις μεταξύ Επιτροπής ε, και κρατών μελών, δηλαδή που αφορά τις χώρες δικαιούχους για να ορίσουμε καλύτερα την ε, πολιτική συνοχή στα εδάφη μας. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση επιτροπής ε, τα επόμενα, τους επόμενους έξι μήνες έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη διαχείριση και τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις πόλεις που θα είναι οι νέοι πρωταγωνιστές ε, τα επόμενα έξι χρόνια αυτής της πολιτικής έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε σχέση με συμφωνίες, εταιρικέ συμφωνίες που να είναι δυναμικές και να μπορούν να ενταχθούν στην πολιτική συνοχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκοτσολίνο, τον συνάδελφό μου από την ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών. Ξέρω ε, πόσο έχει ασχοληθεί για την προώθηση των πόλεων και ο ρόλος των πόλεων ε, θα πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα διότι εντάσσονται στις περιφέρειες ε, και όπου διαμένει το 75% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ρυθμιστικό πλαίσιο που ήδη έχει εγκριθεί. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε μια συλλογική διαδικασία όπου συμμετέχουν οι τροπικές, οι περιφερειακές αρχές και η ΜΚΟ καθώς και η κοινωνία των πολιτών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι ξέρω από τις συζητήσεις ότι δεν εγκρίναμε αυτή την αρχή μόνο για να υπάρχει κάτι επιχάρτου αλλά επειδή θέλουμε οι δικαιούχοι αυτών των επενδύσεων να λαμβάνουν απτές αποφάσεις. Ε, ως προς τη διαδικασία γνωρίζετε ότι με αυτόν τον κανονισμό έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, έτσι ώστε να προωθήσουμε μια διαδικασία απλούστευσης των κανόν, να χρησιμοποιήσουμε τα ηλεκτρονικά μέσα και επίσης Υπάρχουν κανόνες που θα πρέπει να απλουστευτούν από τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία χρειάζονται 40 υπογραφές ε, για να συναυθεί μια συμφωνία επενδύσεων και αυτό δεν προαπαιτείται από την ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε μια εξισορρόπηση πραγμάτων και σας είπα εξ αρχής ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε κανένα συμβιβασμό σε σχέση με τις πληρωμές, τις υποχρεώσεις και τις πληρωμές. Σας ευχαριστώ. Η συμπληρωματική σας ερώτηση. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αναλάβουμε μία αμοιβαία υποχρέωση, δηλαδή τους επόμενους μήνες μαζί με τα κράτη-μέλη να κωδικοποιήσουμε τους, ε, τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης, τις εταιρικές συμφωνίες, για να δούμε κατά πόσο μπορεί και η Επιτροπή να επανέλθει και να μας ε, μιλήσει για αυτή την εφαρμογή, αυτή η εφαρμογή των εταιρικών σχέσεων. Απάντηση. Η κυρία Κρέτσου. Με μεγάλη χαρά θα προσέλθω ενώπιον σας γιατί πιστεύω ότι οι συμφωνίες ε, εταιρικές σχέσεις που έχουν συναυθεί είναι 16-17 και από όσο γνωρίζω ο Επίτροπος Χαν θα προωθήσει αυτή τη διαδικασία μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Ε, εν πάση περιπτώσει θα ξεκινήσουμε συζητήσεις για τα επιχειρησιακά προγράμματα, να δούμε τι περιθώρια έχουμε έτσι ώστε να θέσουμε σε εφαρμογή τις εταιρικές συμφωνίες. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Τόμας Πορέμπα. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να, ρωτήσω την... Ε, να θέσω μια ερώτηση εκ μέρους του ECR και καταρχήν θα ήθελα να σας, να σας ζητήσω να μας αναπτύξετε την άποψή σας για την χάραξη μιας μακροοικονομικής στρατηγικής για τα Καρπάθια που είναι μια από τις ε, φτωχότερες ε, ε, περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρείτε ότι τα Καρπάθια χρειάζονται ένα ξεχωριστό φάκελο εντός των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρόκειται ως Επίτροπος να προωθήσετε αυτή την ιδέα, αυτή τη σκέψη. Οι μικρο- και μακροπεριφέρειες ε, είναι ένα αποδοτικό μέσον και γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο μακροπεριφέρειες του Δούναβη και των Βαλτικών χωρών και της Βαλτικής και στη συνέχεια θα προωθήσουμε τα Ιόνια νησιά και την Αδριατική. Ως προς τα Καρπάθια μπορώ να σας πω ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία και εγώ είμαι πολύ κοντά σε αυτή τη συμφωνία όπως μπορείτε να κατανοήσετε και ε, οπωσδήποτε για τη σύσταση μακροπεριφερειών θα πρέπει να αναλάβουν αυτή την δέσμευση τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται κινητοποίηση των κρατών ε, μελών που αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις μέσα στα πλαίσια ενός ε, διαλόγου και πολιτικής θέλησης. Και βεβαίως με βάση τα κονδύλια που έχουμε στη διάθεσή μας και την ε, τρέχουσα νομοθεσία. Σε σχέση με τις μακροπεριφέρειες, νομίζω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν αυτό το διάβημα και να υποβάλουν το αίτημα στο Συμβούλιο. Από την άλλη πλευρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα πρέπει να διευκολύνει τα κράτη-μέλη. Δεν νομίζω από, ότι από τις ε, Βρυξέλλες μπορούμε να διαχειριστούμε τα προβλήματα του Δούναβη, των Καρπαθίων, της Αδυρατικής ή άλλων τμήματων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τοπικές αρχές και οι τοπικοί εταίροι θα πρέπει να ασχοληθούν με τις μακροπεριφέρειες. Θα πρέπει φυσικά να δούμε και τον, την προσθέμενη αξία των μακροπεριφερειών και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για να ε, ορίσουν τις κοινέ προκλήσεις που αφορούν συγκεκριμένες περιφέρειες και να λάβουν και ευθύνες για τις αντίστοιχες περιφέρειες. Εγώ τάσομαι υπέρ της σύστασης μακροπεριφερειών έτσι ώστε να κινητοποιηθούν οι τοπικές αρχές στα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει τα κράτη στο διαβήμα τους αυτό. Ήθελα να σας ζητήσω να τηρείτε το χρόνο. Ε, συμπληρωματική ερώτηση παρακαλώ. Μια δεύτερη σύντομη ερώτηση. Θα ήθελα να μας πείτε την άποψή σας ε, τι λύσεις θα πρέπει να εφαρμοστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι διαφορές στην ανάπτυξη των περιφερειών. Πώς ε, πρόκειται να εξασφαλίσετε ότι το δυναμικό των περιφερειών θα μπορέσει να αποδώσει καλύτερα, να αξιοποιηθεί καλύτερα και να, ούτως ώστε να δημιουργήσει οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής. Παρακαλώ, η Επίτροπος. Είναι γεγονός ότι θα πρέπει να μειωθούν οι οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές διαφορές. Αυτό είναι απότερο στόχος της περιφερειακής πολιτικής και έμπρακτα αποτελεί υποχρέωσή μας να συνεισφέρουμε μαζί με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να μειώσουμε αυτό το χάσμα και γι' αυτό οι πλέον αναπτυγμένες περιφέρειες ε, λαμβάνουν το 80%. Γι' αυτό έλεγα ότι θα πρέπει να γίνει μία διαφοροποίηση και είπα στην βασική μου εισήγηση ότι αυτές οι χώρες που λαμβάνουν ένα τόσο υψηλό ποσοστό των ταμείων ε, αφορούν ε, περιφέρειες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο. Γι' αυτό θα πρέπει να καταβάλουν ε, προσπάθεια για να βελτιστοποιήσουν την πολιτική συνοχή, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, γιατί θα πρέπει να προωθήσουμε την ε, αρμονική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να υπάρξει μια εξισορρόπηση και μείωση αυτού του χάσματος. Γι' αυτό αποτελεί μέλημά μας να εφαρμόσουμε τους κανονισμούς σωστά λαμβάνοντας υπόψη τις ε, προτεραιότητες έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα χρηματοοικονομικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές ε, τις, ε, αυτά τα μέσα που τους ε, προσφέρουν, προσφέρει το ρυθμιστικό πλαίσιο, γιατί στην περίοδο αυτή κρίσης είναι ύψη της σημασίας να μπορέσουμε να δείξουμε την αλληλεγγύη μας για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχετε μόνο ένα λεπτό σας υπενθυμίζω στην απάντηση για την απάντηση στην συμπληρωματική ερώτηση. Ο κύριος Γιάκοφτσίτς. Καλώς ορίσατε. Εξ ονόματος των μελών ε, της ομάδας των φιλελευθέρων, Άλντε. Για το μέλλον της πολιτικής συνοχής μετά το 2020 είναι σημαντικό να μειωθεί και το ποσοστό σφαλμάτων για να αποφευθούν και μελλοντικέ περικοπές του προϋπολογισμού. Ποια μέτρα μπορείτε να θεσπίσετε ώστε οι χώρες μέλη να λάβουν πιο σοβαρά υπόψη τους το καθήκον ελέγχου. Διότι το ελεγκτικό συνέδριο λέει ότι 50% των σφαλμάτων θα έπρεπε να είχαν ήδη εντοπιστεί από τις ελεγκτικές αρχές των χωρών μελών. Και τι πολιτική θα αναλάβετε στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής για την περιφέρεια της Αδριατικής και σε σχέση με τη διεύρυνση μελλοντικά της Ευρώπης προς νότια-ανατολικά. Δύο λεπτά παρακαλώ κυρία υποψηφία. Όπως είπα και στην αρχή, θα γίνει αυτή η αποτίμηση απόδοσης για την περίοδο μετά το 2020 και θα θέλαμε τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήδη από την αρχική φάση για να συζητήσουμε τη βελτίωση των κανονισμών. Θα πρέπει να δώσουμε μάχη για τον προϋπολογισμό για την περίοδο μετά το 2020. Όλα αυτά θα γίνουν λαμβάνοντας υπόψη μια σαφή ανάλυση που θα γίνει από κοινού του αντικτύπου των μέτρων σε σχέση με την απλούστευση, την αιρεσιμότητα εξάντε... και τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης για την χρήση όλων των χρηματοοικονομικών και εδαφικών μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας Νομίζω ότι θα έρθει η στιγμή να γίνει αυτή η ανάλυση, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, διότι η στρατηγική του 2020 και μετά το 2020 θα πρέπει να δημιουργήσει απασχόληση και ανάπτυξη. Και επειδή και εγώ προέρχομαι από αυτή την περιφέρεια, κατανοώ το ερώτημά σας σε σχέση με την ανάπτυξη αυτών των περιοχών. Νομίζω ότι σε αυτά τα πλαίσια η περιφερειακή πολιτική αποκτά μεγαλύτερη σημασία διότι είναι το μόνο μέσο να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες να αναπτυχθούν. Υπάρχουν χώρες μη μέλη που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των στρατηγικών και θέλουμε να βοηθήσουμε για την σταθερότητα σε αυτές τις χώρες και για την ασφάλεια των συνόρων μας. Θέλουμε λοιπόν να χορηγήσουμε βοήθεια σε αυτές τις χώρες έτσι ώστε ίσως και το 2019 η εν λόγω χώρα να μπορέσει να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επερώτηση. Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να συνδυάσουμε τις διάφορες πολιτικές για να σταθεροποιήσουμε περισσότερο την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έχω όμως και άλλη μια ερώτηση. Θα ζητήσετε από τις υπηρεσίες σας να κάνουν περισσότερους ελέγχους απόδοσης ώστε να στοχεύσουν περισσότερο στην αποδοτικότητα της πολιτικής συνοχής και πώς θα ε, αναπτύξει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικούς της ελέγχους βασισμένους στο κίνδυνο, risk-based audits. Αυτή η δραστηριότητα ελέγχου έχει μεγάλη σημασία διότι όπως σας είπα κάθε ευρώ του προϋπολογισμού θα πρέπει να δαπανηθεί σωστά και θα πρέπει να βελτιστοποιήσουμε την ε, απόδοση των χρημάτων αυτή την περίοδο γίνονται πολλοί έλεγχοι και ξέρετε ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να εγγυηθεί, να προβάλλει εγγυήσεις ήδη από την αρχή του κάθε οικονομικού έτους. Εάν υπάρχουν υποψίες, τότε άλλες ελεγκτικές αρχές θα πρέπει να προβούν στην επαλήθευση όλων των δράσεων που αφορούν την καταβολή χρημάτων. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι όταν υπάρχουν σοβαρές περιπτώσεις η Όλαφ αναλαμβάνει την, τον έλεγχο. Άρα θα συνεργαστούμε και με την ε, Όλαφ. Δεν έχω, ε, δεν έχω απαντήσει σε σχέση με τα σφάλματα που αναφέρεται. Θα τα δω στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και των ελέγχων. Ευχαριστούμε και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Μαριέ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κρετού εκ μέρους της, ε, των μελών της ΚΟΕ, NGL. Καλώς ήρθατε. Το θέμα των 23 δις αναφέρθηκε, δεν θα επανέλθω, παρόλο που μας ανησυχεί πολύ, γιατί προσβάλλει την ίδια την αξιοπιστία της περιφερειακής πολιτικής και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ίσως πιο σοβαρό ακόμα είναι το εξή. Γνωρίζετε ορισμένε χώρες μέλη αναμένουν να ξαναγίνει η συζήτηση για το ΣΕΦΜΠΕ για να προκειμένου να γίνουν κάποιες περικοπές στον προπολογισμό και αυτό με το κίνδυνο να καταφερθεί ένα σημαντικό πλήγμα στην περιφερειακή πολιτική. Ε, μπορούμε να έχουμε εκ μέρους σας τη δέσμευση ότι θα συνεργαστούμε για να αποφύγουμε την εξέλιξη αυτού του σενάριου. Γνωρίζετε ότι η πολιτική, το μέλλον της ε, περιφερειακής πολιτικής δεν είναι εξασφαλισμένο και πραγματικά καθίστε ιδιαίτερη ευάλωτη συνεπία της κριτικής που ασκεί το ελεγκτικό συνέδριο. Ποια είναι τα μέτρα που θα λάβετε για την ε, πάταξη της απάτης. Să fiu sinceră, Για να είμαι ειλικρινής, περίμενα να μου μιλήσετε για τις πλέον απομακρυσμένες περιοχές, γιατί διάβασα την έκθεσή σας και ε, εντυπωσιάστηκα από το μέλημά σας για αυτές τις απομακρυσμένες περιφέρειες. Σε σχέση με το ερώτημά σας, δεν νομίζω ότι μπορούμε να θέσουμε ένα αμφιβόλο το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο συζητήθηκε μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και θα πρέπει να διατηρήσουμε να τηρήσουμε το νυν νομοθετικό πλαίσιο. Θα πρόκειται για μια κοινή μάχη γιατί θα, δεν θέλουμε να μειωθεί ο προϋπολογισμός. Μπορείτε να βασιστείτε σε μένα. Όπως γνωρίζετε και όπως είπε και ο κύριος Βανίστελ Ρόι, δεν είμαι εμπειρογνώμων, προετοιμάστηκα για αυτή την ακρόαση και κατά τη διάρκεια της εργασίας μου θα βελτιώσω αυτό το πλαίσιο διότι η περιφερειακή ανάπτυξη είναι ύψης της σημασίας και ξέρουμε παράλληλα ότι πολλοί επιτίθενται στις περιφέρειες και θέλουν να μειώσουν τα κονδύλια για την περιφερειακή ανάπτυξη. Θα πρόκειται για μια κοινή μάχη που θα δώσουμε και θα ήθελα να είσαστε σύμμαχοί μου, διότι γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα με υποστηρίξει. Θα πάω με άλλον αέρα αν θέλετε, αν ξέρω ότι έχω την υποστήριξή σας. Και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μας ε, ακολουθήσει. Δεν θα πρέπει να δεχτούμε μειώσεις. Αυτή είναι η μοναδική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτική επενδύσεων που οδηγεί σε απτά αποτελέσματα και οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Επερώτηση. Στο μια συμπληρωματική ερώτηση για τις απομακρυσμένες περιφέρειες οι περιφέρειες αυτές έχουν αναγνωριστεί στο πλαίσιο της συνθήκης από ένα άρθρο, από το άρθρο 349. Και το άρθρο αυτό... Ε, και ε, αναφέρονται λοιπόν σε αυτό το άρθρο τι πρωτοβουλίες προτίθεστε εσείς να πάρετε ούτω ώστε το άρθρο αυτό να εφαρμοστεί πλήρως στο σύνολο των ευρωπαϊκών πολιτικών ε, και κυρίως εκ μέρους των του συνόλου των επιτρόπων. Γνωρίζετε το Κοινοβούλιο ενέκρινε στην αρχή της έκθεσης μια έκθεση πρωτοβουλίας για τις εξόχους απόκεντρες ε, ε, περιφέρειες, περιοχές και ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που πρόκειται να λάβετε ούτω ώστε τα μέτρα που προτείνει η έκθεση αυτή να μπορέσουν να εφαρμοστούν. Ευχαριστώ, έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σας. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Όπως ξέρετε, οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες έχουν ένα ειδικό καθεστώς γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις επειδή γεωγραφικά είναι απομακρυσμένες από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Γι' αυτό θα πρέπει να προσδώσουμε μεγάλη σημασία για την τήρηση των άρθρων που προαναφέρατε και για να βοηθήσουμε αυτές τις ε, περιφέρειες, τις πλέον απομακρυσμένες. Εάν διοριστώ, θα είμαι επίτροπος όλων των ε, περιφερειών. Παράλληλα, θεωρώ ότι λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη πόρων ε, πρέπει να τύχουν και μεγαλύτερη σημασία. Θα μεταβώ σε αυτές τις περιφερειές για να δω επιτόπου ποιες είναι οι ανάγκες αυτών των περιφερειών γιατί θεωρώ ότι αποτελούν μοναδική αξία ανοίγματο της Ευρώπης προς τον κόσμο και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ενιαία ανάπτυξη. Νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε με τον πρόεδρο Γιούνκερ και με τον επίτροπο Κατάινεν που θα είναι υπεύθυνο για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και με την Πορτογαλία, Γαλλία και Ισπανία καθώς και με τους κυβερνώντες αυτών των ε, απομακρυσμένων ε, περιφερειών χρειάζεται ανταλλαγή απόψεων. Εσείς ξέρετε άμεσα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι περιφέρειες και θα πρέπει να εξεύρουμε λύσεις από κοινού μέσα στα πλαίσια μιας ενιαίας ε, στρατηγικής για τις πλέον απομακρυσμένες περιφέρειες, λαμβάνοντας υπόψη την ολοκλήρωσή τους. Σας ευχαριστώ. Θα ακολουθήσει η κυρία Βάνα. Καλημέρα κυρία Κρέτσου, εξ ονόματος των Πρασίνων. Η σημασία του ρόλου των αστικών κέντρων στην πολιτική συνοχή ήδη αναφέρθηκε προηγουμένως, διότι τα αστικά κέντρα είναι και μοχλός ανάπτυξης, αλλά και προσφέρουν υπηρεσίες και σε όλη την περιφέρεια και ειδικότερα για την επίτευξη των στόχων 2020. Τώρα οι πόλεις και τα άλλα κέντρα έχουν ανάγκη από επενδύσεις, για παράδειγμα για την προστασία του κλίματος, για την απασχόληση, για την καταπολέμηση της φτώχειας. Και οι επενδύσεις αυτές δεν είναι πλέον επαρκείς, διότι αναγκάστηκαν και οι πόλεις, και οι δήμοι, να περικόψουν και αυτοί τους προϋπολογισμούς τους. Ερώτηση. Πώς θα εξασφαλίσετε ή πώς θα συμβάλλει συγκεκριμένα η πολιτική συνοχή, έτσι ώστε οι πόλεις στο μέλλον και διαρθρωτικά αλλά και λειτουργικά να μπορέσουν να παραμείνουν σε, να έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτούν σε επαραδίτες αυτές τις επενδύσεις. Ευχαριστώ. Παρακαλώ δύο λεπτά. Όπως προείπα, κατά την άποψή μου, οι πόλη θα είναι ο φυσικός εταίρος της Επιτροπής διότι εκεί βρίσκεται το 75% του ευρωπαϊκού πληθυσμού και όπως είπατε και εσείς, διανοίγονται άλλοι, άλλες οδοί ανάπτυξης και έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις που σχετίζονται ιδιαίτερα με τον κοινωνικό αποκλεισμό. Θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς. Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί ένα από τα 11 σημεία που εγκρίναμε στη νέα μας αναθεωρημένη πολιτική. Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα προς αυτό το τομέα. Και υπάρχει και ένα θέμα επικοινωνίας που θα πρέπει να προωθήσουμε. Δηλαδή δεν θα πρέπει να μας απασχολεί μόνο η οικονομική ανάπτυξη και η απασχόληση, αλλά να μην αφήσουμε κανέναν πίσω. Δηλαδή το θέμα της στέγης και της κοινωνικής στέγης και στέγασης είναι ύψης της σημασίας. Έτσι πρέπει να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους. Από όσο γνωρίζω από τους ε, υπολογισμούς, 5,2 δις ευρώ θα δοθούν για την στέγη, για τη στέγαση των κοινωνικών αποκλεισμένων και για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Ξέρετε ότι έχουν γίνει πολλές ε, κοινωνικές ε, επενδύσεις, κοινωνικού χαρακτήρα, ηλεκτροδότηση στέγης και υποστήριξη αυτής της ευάλωτης κατηγορίας ανθρώπων για να, μπορέσει, να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να επιβιώσουν καλύτερα. Και αυτό το είδαμε στα πλαίσια του προγράμματος 2007-2014 πληρωματική σας ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κρέτου για αυτή την απάντηση. Εσείς αναφερθήκατε ίδια στην, ε, στο σημαντικό ρόλο των δημόσιων υπηρεσιών όσον αφορά την επαρχή υπηρεσιών για τις πόλεις. Και στη Λευκή Βίβλο ε, της Κομισιόν του 2008 αναφέρεται ο σκοπός κοινή ε, της ε, περιφερειακής πολιτικής να υπάρχει πρόσβαση στις δημόσιες αυτές υπηρεσίες. Αυτή η διάσταση δεν αναφέρεται στην έκτη έκθεση συνοχής, δεν αναφέρονται αυτές οι δημόσιες υπηρεσίες και συνήθως ε, υπάρχουν κάποιες ε, τάσεις απελευθέρωσης σε αυτό το τομέα και ιδιωτικοποίηση για τις υπηρεσίες κοινή ωφέλειας. Ε, πώς θέλετε να εξασφαλίσετε ότι οι υπηρεσίες κοινή ωφελίας αναφέρατε τη στέγαση, την εκπαίδευση, την υγεία, την υδροδότηση κλπ. να μην συρρυκνωθούν και το δημόσιο να συνεχίζει να εξασφαλίζει αυτές τις υπηρεσίες κοινή ωφέλειας στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Ευχαριστώ. Έχετε ένα λεπτό για να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Όπως σας είπα... Οι υπηρεσίες κοινή ωφελία διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθούν. Αποτελούν κοινή αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρονται στη συνθήκη και στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινή ωφελίας που προωθούν την κοινωνική και εδαφική συνοχή θα πρέπει να έχουμε μια πιο γενναιόδορη πολιτική ως προς αυτές τις υπηρεσίες που αφορούν την εκπαίδευση, την υγεία, την περίθαλψη των παιδιών, την κοινωνική περίθαλψη και το θέμα της στέγασης των ευάλωτων κατηγοριών. Όλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες και έτσι μπορεί να γίνει πιο δελεαστική και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία συγχρηματοδότησης αυτών των ε, υπηρεσιών, ιδιαίτερα στους τομείς ε, της υγείας, της εκπαίδευσης, της ε, μεταφοράς, της απομάκρυσης των αποβλήτων και της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Ευχαριστώ. Now, η πρόεδρος. Ευχαριστώ. Η κυρία Νταμάτο. Καλημέρα σας και καλώς ορίσατε. Η πολιτική συνοχή μέσα στα πλαίσια της αιρεσιμότητας έχει πολλά προβλήματα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η οικονομική διακυβέρνηση. Σήμερα η, οικονομική διακυβέρνηση δεν λαμβάνει υπόψη ότι η πολιτική ε, συνοχή θα έπρεπε να εκπροσωπεί πάνω από το 50% των δημόσιων επενδύσεων. Τα ταμεία επέτρεψαν τις επενδύσεις στο δημόσια και ιδιωτικό τομέα, όπως δείχνει και μια μελέτη Ρέτζι. Υπάρχουν περιφέρειες όμως που αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις οικονομικές και κοινωνικές. Δυστυχώς υπάρχει προσέγγιση top-down και όχι top-up. Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη όλες τις συνέργειες όλων των οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων έτσι ώστε οι περιφέρειες να μην υποστούν τις συνέπειες των, ε, των μεγάλων δημοκρατικών ε, και κοινωνικών ελλημάτων των κρατών μελών. Δύο λεπτά για να, Δύο για να απαντήσετε παρακαλώ. Όπως είπατε υπάρχει αυτό το ζήτημα, το γεγονός ότι ορισμένα κράτη-μέλη δεν μπορούν να απορροφήσουν ούτε το 50% αυτών που, των πόρων που έλαβαν ε, το, από το 2007 μέχρι το 2013, ιδιαίτερα τα νέα κράτη-μέλη. Νομίζω όμως ότι βελτιώθηκε η κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι ε, η Επιτροπή έχει χρέος να βοηθήσει αυτά τα κράτη να διαχειριστούν καλύτερα την κατάσταση γιατί σας είπα ότι αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό ακόμα και από τα χρήματα, δηλαδή η διαχείρισή τους, διότι τα περισσότερα σφάλματα, και επανέρχομαι στις προγενέστερες ερωτήσεις, αφορούν την κακοδιαχείριση. Γι' αυτό νομίζω ότι με τις ε, ρυθμιστικές απλουστεύσεις θα φτάσουμε σε αυτά αποτελέσματα, ορίζοντας τις βασικές προτεραιότητες ανάπτυξης και μία αλλαγή σε αυτές τις περιφέρειες. Γνωρίζω ότι προέρχεστε από μία περιφέρεια που έχει πληγεί ιδιαίτερα από τη Σικελία και θα ήθελα να σας εκφράσω την αλληλεγγύη μου. Ε, δεν θα πρέπει να πλήτεστε από την ε, κακοδιαχείριση. Η μακροαιρεσιμότητα εγκρίθηκε από εσάς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, διότι ε, αντλήσαμε από τα διδάγματα μάλλον από την κρίση και γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να γίνουν εύρωστες επενδύσεις έτσι ώστε να μην διασπαθιστεί το δημόσιο χρήμα. Άρα αυτές οι συνθήκες της μακροαιρεσιμότητας έχουν μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι αναφέρεστε στο τελευταίο μέτρο αναστολής πληρωμών. Αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήξει, γιατί αποτελεί το πέρας μιας διαδικασίας όπου το κράτος πληροφορείται και επιπλήτεται διότι πρέπει να προβεί σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Θα επεκταθώ όταν θα έχω την ευκαιρία. Μία επερώτηση τώρα που αφορά την οικονομική πτυχή. Δηλαδή το περιφερειακό ΑΕΠ που είναι βασικός δείκτης για την επιλεξιμότητα και για να δούμε ποιες θα είναι οι ποσοστώσεις χρηματοδότησης στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές. Αυτό είναι μία λανθασμένη προσέγγιση, γιατί ο δείκτης output όπως αυτός του ΑΕΠ είναι κάτι το ανεπαρκές. Χρειάζονται περισσότερα εδαφικά κριτήρια πρόσφατες στατιστικές ε, για να δούμε ποιες είναι οι εδαφικές ε, ιδιαιτερότητες. Θα μπορέσετε να αναθεωρήσετε άρδιν αυτή την πολιτική συνοχής έτσι ώστε τα κονδύλια να διανέμονται σωστά και να μην χρησιμοποιείτε ως μοναδικό κριτήριο το ΑΕΠ. Η πρόεδρο. ένα λεπτό. Ε, σίγουρα και φυσικά γίνεται αυτή η συζήτηση για αυτό το κριτήριο, αυτό το δίκτυ και τη χρήση του και μπορώ να σας πω ότι το μοναδικό κριτήριο που έγινε αποδεκτό ομόφωνα είναι το ανακεφαλή ΑΕΠ. Όπως γνωρίζετε λαμβάνουμε υπόψη το ανακεφαλή ΑΕΠ που είναι κάτω από το 75% του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Θα πρέπει ε, εμείς να δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε εμείς. Στο Συμβούλιο θα πρέπει να γίνουν συζητήσεις σε σχέση με το κριτήριο αυτό. Νομίζω ότι έχετε δίκιο τα κονδύλια θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανθρώπινες ανάγκες. Γι' αυτό υπάρχει και η εταιρική αυτή αρχή. Έτσι ώστε να έχουμε την συμμετοχή και των τοπικών αρχών της κοινωνίας των πολιτών για να μας πούν ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες αυτών των πολιτών. Και ξέρω ότι υπάρχουν χώρες όπου αυτή η αρχή δεν εφαρμόζεται όπως πρέπει, διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε διαφορετικές πολιτισμικές βάσεις, υπάρχουν χώρες με μεγαλύτερη συγκεντρωτική διακυβέρνηση και γι' αυτό θα πρέπει να ορίσουμε από κοινού ένα ενιαίο πλαίσιο. Νομίζω λοιπόν ότι οι νέοι κανονισμοί θα πρέπει να εφαρμοστούν από όλα τα κράτη-μέλη και περιφέρειες έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στους απότερους ε, στόχους των περιφερειών. Thank you. Now begin our... Ευχαριστώ. Θα, θα αρχίσουμε τώρα τον δεύτερο γύρο των ερωτήσεων. Εδώ επιθυμώ να σας υπενθυμίσω ότι έχετε τρία λεπτά, συγγνώμη, τρία λεπτά ένα λεπτό ερώτηση, δύο λεπτά απάντηση. Ήδη έχουμε ξεπεράσει κατά 10 λεπτά το χρονοδιάγραμμά μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν με τον κύριο Ντόιτς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, θεωρείτε ότι όπως κάναμε το 2000-2006 αν θεωρείται το 2007 έως 2013, μια παράταση της ίδιας περίοδου, γιατί όπως είπε και ο κ. Χάν, ελπίζει ότι μέχρι τέλους του έτους 100 επιχειρησιακά προγράμματα θα μπορέσουν να έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βρισκόμαστε όμως πολύ μακριά ακόμα από αυτό το στόχο. Και Ούτως ή άλλως έχουν σχεδιάσει 460 τέτοια προγράμματα ή έργα ή χώρες μέλη. Έχετε πρόθεση να επιταχύνετε τη διαδικασία έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όπως είπατε και εσείς, είναι πάνω από 23,4 δισεκατομμύρια το έλλειμμα των πληρωμών και η περίοδος των λογαριασμών, εφόσον παραταθεί από πληρωμή των λογαριασμών δηλαδή, θα μειώσει την πίεση. Αν δηλαδή προτίθεστε να παρατείνετε τις προθεσμίες αποπληρωμής, όπως είχατε κάνει και στην προηγούμενη περίοδο, αν θα το κάνετε και τώρα. Δύο λεπτά για να απαντήσετε. Uh, uh, Γνωρίζω ότι υπάρχει αυτό το αίτημα παρέκτασης αυτής της περίοδου μέχρι και το τέλος του 2015 και αργότερα. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία δεν αποπλήρωσαν τα ποσά αυτά για την περίοδο 2007-2013 έχουν να πληρώσουν ένα 15%, 20%. Θα πρέπει να τα βοηθήσουμε έτσι ώστε το 2015 να βρουν το καλύτερο ε, τρόπο αποπληρωμής. Θα ήθελα να σας πω ότι κατά την άποψή μου δεν θα πρέπει να θυσιάσουμε την ποιότητα των προγραμμάτων για λόγους απορρόφησης ε, και μόνο. Αυτά είναι ποιοτικά προγράμματα και αν είναι πράγματα ποιοτικά, πράγματι ποιοτικά και ανταποκρίνονται στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, θα πρέπει να τηρηθούν Δηλαδή με ανησυχεί αυτό το κριτήριο της ταχύτητας. Δηλαδή ας αφήσουμε την ε, ποιότητα στην άκρη για να δείξουμε ότι καταβάλουμε τα χρήματα το συντομότερο δυνατόν. Καταρχήν θα πρέπει να έχουμε αποτελέσματα. Γι' αυτό θα πρέπει από κοινού να δούμε μαζί με το Συμβούλιο ποια, ποιες είναι οι δυνατότητες γιατί ξέρω ότι και η Ιταλική Προεδρία ζήτησε την ε, παράταση αυτής της περίοδου, αλλά θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε αποδοτικά τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι το τέλος του 2015. Και παράλληλα θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας για τα επιχειρησιακά προγράμματα έτσι ώστε να τεθούν σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν για την περίοδο 14-20. Ο κύριος Βόν. Καλημέρα, κύριε Κρέτσου. Το Κοινοβούλιο υποστήριξε τη δημιουργία νέων μηχανισμών community-led, ε, local development, κοινά προγράμματα ολοκληρωμένες περιφερειακές επενδύσεις, έτσι ώστε να υπάρξει και μια εκ των κάτω προσπάθεια εξασφάλισης της συνοχής. Ερώτηση λοιπόν, ως Επίτροπος θα λάβετε μέτρα αξιολόγησης της χρήσης αυτών των νέων μηχανισμών. Δεύτερο, ως Επίτροπος θα εξετάσετε εάν οι συμφωνίες συνεργασίας χωρών μελών πραγματικά έχουν οδηγήσει σε συνεργασία και με άλλους stakeholder. Ευχαριστώ. Παρακαλώ δύο λεπτά για να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Όπως γνωρίζετε, στην περιφερειακή πολιτική η εδαφική ενότητα και οι εδαφικές μονάδες έχουν πολύ μεγάλη σημασία και σας ευχαριστώ για τα νέα αυτά εδαφικά μέσα που προβάλλεται πρόκειται για ολοκληρωμένες επενδύσεις και την τοπική ανάπτυξη υπό την ευθύνη της Ευρωπαϊκής, της Ένωσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι αυτή η μετάβαση αρμοδιοτήτων προς τις περιφερειακές αρχές οδηγεί στην ανάθεση ευθυνών και σε τοπικό επίπεδο έτσι ώστε τα κονδύλια να βρίσκονται πιο κοντά στον πολίτη. Πρόκειται για απαράβατο όρο στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση αυτών των μέσων, διότι η αρχή της επικουρικότητας θα πρέπει να τηρηθεί αλλά η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση πολύ συχνά οδήγησε σε αρνητικά αποτελέσματα. Πρόκειται όμως για ένα επιπρόσθετο στοιχείο το οποίο σε τελευταία ανάλυση θα βελτιώσει τον τρόπο λήψης αποφάσεων. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να γνωρίζουν πολύ καλά τους νέους κανονισμούς οι οποίοι εγκρίθηκαν και σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσουν μεγάλη σημασία σε αυτά τα μέσα, σύμφωνα με την πρόοδο που έχει επιτελεστεί στα κράτη-μέλη ε, ως προς τη χρήση αυτών των μέσων. Ευχαριστώ. Κύριος Πόλτσακ. Κυρία Κρέτσου, έχω την εξής ερώτηση συμμετοχή των τοπικών εταίρων, οργανώσεων πολιτών κλπ. Στην δημιουργία για τη διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτικών. Αυτό παραμένει υποχρεωτικό μέρος των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την ε, Περιφερική Ανάπτυξη και θα είναι και δυνητικό για ορισμένα άλλα ταμεία, όπως το Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Θάλασσας και Αλίας. Η μέθοδος αυτή έχει διευρυνθεί πολύ. Αυτό είναι αναμφίβολο. Χρησιμοποιείται η μέθοδος αυτή ωστόσο πλήρως. Υπάρχει χώρος βελτίωσης. Υπάρχει λόγος να θεωρήσει κανείς ότι η προσέγγιση ELD είναι πλέον ξεπερασμένη. Thank you. You have minutes to answer the question. Παρακαλώ απαντήστε σε δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Όπως σας είπα, αυτά τα μέσα που σχετίζονται με το, την αρχή Community Led Local Development σχετίζονται με την προώθηση της τοπικής συνεργασίας έτσι ώστε οι τοπικές αρχές να ασχοληθούν με την ανάπτυξη της εκάστοτε περιφέρειας. Πρόκειται για τα διδάγματα που αντλήσαμε από το πρόγραμμα LEADER, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ε, σε ευρία κλίμακα πάνω από 20 χρόνια και προσέδωσε μεγάλα και σοβαρά αποτελέσματα. Ε, διαμέσου αυτής της αρχής ε, προωθούμε μια πολιτική συνοχής και ενδυνάμωσης ενίσχυσης των ε, τοπικών κοινοτήτων. Αυτό αποτελεί ένα μεγάλο κέρδος για την ανάπτυξη των αγροτικών περιφερειών ιδιαίτερα. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι βασικές ανάγκες των αγροτικών περιοχών και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε αξιολογήσεις για να δούμε πόσο τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μέσα έτσι ώστε να εκπροσωπηθούν όλοι οι τομείς ε, της ε, κοινωνίας και νομίζω ότι οι τοπικές και περιφερικές αρχές φέρουν μεγάλη ευθύνη και θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους τοπικούς παράγοντες και τον επιχειρηματικό κόσμο, έτσι ώστε να συμμετάσχει ενεργά ε, σε, αυτό, αυτή την περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της επικουρικότητας. Ευχαριστώ και ακολουθεί η ερώτηση του κ. Μποστινάρου. Καλώς ήρθατε κυρία υποψηφία επίτροπε και συνεχίζω στα αγγλικά. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω απέναντί μου την υποψήφια επίτροπο από τη χώρα μου. Ε, ωστόσο εδώ θα μιλήσουμε για την Ένωση. Σημαντικό μέρος του Ταμείου Συνοχής 10 από 66 δισεκατομμύρια λοιπόν μετά, ε, ε, ε, ευρώ μπαίνουν στο νέο εργαλείο διευκόλυνσης της ε, συνδέοντας την Ευρώπη, την νέα διευκόλυνση. Αυτή η διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη και η διαδικασία επιλογής γίνονται στις Βρυξέλλες και όχι στο εθνικό επίπεδο. Αποφασίστηκε μετά από αγώνα της παρούσας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με συμμετοχή όλων των συναδέλφων μου. Καταφέραμε λοιπόν να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατηρήσει τα χρήματα στα, στους εθνικούς φακέλους μέχρι το 2016. Η ερώτησή μου προς εσάς έχει ως εξής. Ποια μέτρα θεωρείτε ότι πρέπει να λάβουν οι χώρες μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξασφαλιστεί ότι οι χώρες μέλη που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν τις χέρειες θα μπορέσουν ωστόσο να υποφεληθούν πλήρως από την διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη και να χρηματοδοτήσουν έτσι έργα ποιότητος. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη συμμετοχή σας σε αυτό τον μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη. Ξέρω ότι διαδραματίσατε σημαντικό ρόλο και εάν διοριστώ θα συνεργαστούμε πολύ καλά. Όπως είπατε, ο μηχανισμός συνδέοντας την Ευρώπη είναι ένας μηχανισμός ύψης της σημασίας διότι έχει άμεση σχέση με το τομέα της ενέργειας και των μεταφορών και προτίθεται να καλύψει κενά στα επιχειρησιακά προγράμματα. Όπως είπατε, τα ταμεία συνοχής είναι πολύ σημαντικά μέσω της μεταφοράς κονδυλίων στο μέσο αυτό, συνδέοντας την Ευρώπη. Χρέος μου λοιπόν θα είναι να συνεργαστώ με την Γενική Διεύθυνση Μεταφορών ιδιαίτερα, έτσι ώστε να προωθήσουμε ποιοτικά προγράμματα μέχρι το τέλος του 2016 για να μην χαθούν αυτά τα χρήματα και θα ενθαρρύνουμε την χρήση αυτών των μέτρων, ιδιαίτερα το ΓΙΑΣΠΕΡΣ που είναι ένα πρόγραμμα της ΕΤΕ για την προετοιμασία μεγάλων προγραμμάτων και αυτά τα προγράμματα μεταφορών και ενέργειας είναι στρατηγικής σημασίας και θα τα παρακολουθήσουμε με μεγάλη προσοχή. Α, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε με περιορισμένους πόρους την πρόθεση αυτών των προγραμμάτων γιατί θα συμπληρώσουν τις ελλείψεις των εθνικών προγραμμάτων όσον αφορά την ενέργεια και τις μεταφορές. κύριος ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, κυρία Υποψήφια, υποψήφια Επίτροπε, θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη δέσμευση που αναλάβατε να συνεργαστείτε στενά με αυτή την Επιτροπή και να την ενημερώνετε. Ε, νομίζω ότι είναι μια φυσική δέσμευση για κάποιον που ήδη έχει εργαστεί επί 8 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά θέλω να εξασφαλίσω ότι θα λησμονήσετε αυτή τη δέσμευση. Μία από τις προτεραιότητες του ΕΛΚ σε αυτή την Επιτροπή είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση. Και ξέρετε ότι έχουμε το οργανισμό για τις κοινέ διατάξεις που εισάγει το πλαίσιο της κοινή στρατηγικής και τις κατευθυντήριες γραμμές για την ολοκληρωμένη εδαφική ολοκλήρωση με τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων. Στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης η ολοκληρωμένη προσέγγιση προβλέπεται ε, αλλά δεν καλύπτεται από τις αποφάσεις της Επιτροπής εκτός ε, εάν ε, δεν εκπληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια θα είναι η δική σας προσέγγιση ούτως ώστε να ενισχύσετε, να θαρρύνετε την αποτελεσματική χρήση της εδαφικής προσέγγισης για την περιφερειακή ολοκλήρωση. Ευχαριστούμε. Έχετε δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Βίγκλερ. Όπως σας είπα, και όπως είπατε και εσείς, θα πρέπει να εξεύρουμε εταίρους πρωτίστως. Ξέρω ότι τα μέλη αυτής της Επιτροπής έχουν μεγάλη πείρα ως προς την περιφερειακή ανάπτυξη. Θα ανταλλάξουμε πληροφορίες και θα είμαι παρούσα στις συζητήσεις της Επιτροπής. Όσον αφορά το ερώτημά σας και σε σχέση με την ε, προσέγγιση το, της ολοκλήρωσης, η περιφερειακή ανάπτυξη έχει επιπτώσει σε πολλούς τομείς, όπως σας είπα στην αρχή, στην καινοτομία, στην έρευνα, στην ενέργεια, στην ψηφιακή ανάπτυξη και έχει μεγάλη σημασία για εμάς να συνεργαστούμε με όλες τις συνιστώσεις για να εξασφαλίσουμε αυτές τις συνέργειες έτσι ώστε τα ταμεία συνοχής να είναι πιο αποτελεσματικά. Θα πρέπει να υπάρχει αλληλοσυσχετισμός των πολιτικών μας. Και ως Επίτροπος, εάν διοριστώ, θα συνεργαστώ για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και θα συνεργαστώ και με άλλους επιτρόπους, τον Επίτροπο Κοινωνικών Εποθέσεων και του Προϋπολογισμού, για να φτάσουμε στους κοινούς μας στόχους δηλαδή την, την ανταπόκριση στο γενικό πρόγραμμα του κυρίου Γιούγκερ. Ευχαριστούμε. Τώρα η ερώτηση του κυρίου Βαν Μίλτεμουρκ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Στα Ολλανδικά. Κυρία Επίτροπε, μιλήσαμε κατά επανάληψη για το ρόλο των πόλεων, ε, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός γιατί γνωρίζετε ότι πάνω από 30% του ευρωπαϊκού πληθυσμού αυτή τη στιγμή διαβιούν σε πόλεις. Το, μέχρι το 2050 θα είναι 80%. Οι πόλεις διδραματίζουν σημαντικό ρόλο για τον κοινωνικό αποκλεισμό ε, και σε άλλα θέματα για την ανάπτυξη κλπ. Και έχουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Έχετε την άποψη ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις ε, πόλεις. Χρειαζόμαστε μια ατζέντα για τις πόλεις. Και τι είδου εργαλεία προτίθεται να δείξετε στο πλαίσιο αυτό. Έχετε σχετικά με τις πόλεις ένα πολιτικό όραμα. Πώς θέλετε να, να ανταποκριθείτε στην, στις ανάγκες ε, των πόλεων. Έχετε δύο λεπτά. Δεν ξέρω κατά πόσο κατάλαβα καλά την ερώτηση. Πρόκειται για τη στρατηγική για τις, για τις αστικές περιφέρειες. Κατάλαβα καλά. It's about urban, urban. Πρόκειται για την, αστικές, την αστική στρατηγική. Στρατηγική για τα αστικά κέντρα, ναι. Σας είπα ότι οι πόλεις αποτελούν μια βασική διάσταση διότι ε, όπως ξέρετε η Γενική Διεύθυνση είναι η Γενική Διεύθυνση για τις Περιφέρειες ε, και τα Μεγάλα Αστικά Κέντρα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει, ε, να συμβαδίζει ο τίτλος του Επιτρόπου με τον τίτλο της Γενικής Διεύθυνσης. γιατί ασχολούμαστε και με τα αστικά κέντρα. Δεν βλέπω λοιπόν γιατί υπάρχει αυτή η ε, διαφοροποίηση της Γενικής Διεύθυνσης από τον τίτλο του Επιτρόπου. Όμως ε, προσδίνουμε μεγάλη σημασία στα αστικά ε, δίκτυα στην Λιψία έχουμε ένα εξαιρετικό σχέδιο, όπως και στη Μάλακα, για τις ιστορικές ε, ζώνες στο Μπρνο, στην Τσεχία. Και θα ήθελα τα κράτη-μέλη να προβούν σε ανταλλαγή απόψεων. Γνωρίζετε επίσης ότι αυτή η δημόσια ατζέντα για τα αριστικά κέντρα έκλεισε την προηγούμενη εβδομάδα και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να φτάσουμε στα σωστά συμπεράσματα και θα πρέπει να αποτανθούμε και στην Επιτροπή Περιφερειών να μας πει ποια είναι η δική της ε, πείρα και θα πρέπει να τηρήσουμε την αρχή της ε, επικουρικότητας. Η επόμενη ερώτηση είναι από την κυρία Μπρέσο. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητή Κορίνα, σε συγχαίρω και εγώ. Ε, η δική σου επιτυχία θα είναι και δική μας. Όταν ε, ε, μίλησε στο Κοινοβούλιο, ο πρόεδρος Γιούνκερ μίλησε για, ε, για ένα τριετές σχέδιο 300 δις ευρώ, μιλώντας για επιπρόσθετα κονδύλια. Πώς μπορούν να ενταχθούν αυτά τα χρήματα στην πολιτική συνοχή μέσα στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής επειδή ε, τα κονδύλια αυτά εγκρίθηκαν, πώς ε, θεωρείτε ότι αυτά τα νέα κονδύλια θα ε, ενταχθούν στις υπάρχουσες πολιτικές για την ενίσχυσή τους. Thank Σας ευχαριστώ και εγώ σας συγχαίρω για ό,τι έχετε επιτύχει στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής. Υπάρχει αυτό το πρόγραμμα που παρουσίασε ο πρόεδρος Γιούνκερ που είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο και είμαι πεπισμένη ότι έχουμε να κάνουμε ένα προϋπολογισμό του ενός τετάρτου του συνολικού προϋπολογισμού για την επιτυχία αυτού του στόχου για την οικονομική ανάπτυξη και την δημιουργική απασχόληση. Υπάρχει αυτός ο κανονισμός και νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια ελιγμού έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε σε αυτή τη φιλόδοξη ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πρόεδρου Γιούνκερ. Ξέρετε ότι ο Πρόεδρος Γιούνκερ μίλησε και για τη χρήση ιδιωτικών πόρων και γι' αυτό θα πρέπει να αλλάξουμε τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε έτσι ώστε να υπάρξει αύξηση επενδύσεων, ιδιαίτερα από τον ιδιωτικό τομέα και νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα χρηματοοικονομικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να ε, έχουμε αυτό το μοχλό και τη δυνατότητα μόχλευσης μέσα στα πλαίσια της ε, καινοτομίας. Μιλάμε για 110 δις ευρώ τα επόμενα χρόνια και θα πρέπει να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ, την ενεργειακή απόδοση και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τις ΜΜΕ και αυτό είναι το βασικό κριτήριο για την εκπλήρωση αυτή του στόχου. Υπάρχουν και άλλα θέματα ε, που αφορούν τον κανονισμό. Δεν μπορώ να επεκταθώ τώρα επί του θέματος. Next Επόμενη ερώτηση από τον κύριο Φίτο. Ε, ε, Σημερίζω με αυτά που είπε η κυρία Μπρέσο. Απλώς θα ήθελα να επεκταθώ λίγο ως προς την ερώτηση. Πολλοί λένε ότι αυτά τα 30 δις ε, δεν μπορούν πραγματικά να είναι επιπρόσθετα. 300 δις, με συγχωρείτε. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ότι αυτά τα κονδύλια αποκλείονται από τα κονδύλια του αρχικού προγραμματισμού. Έχουμε να κάνουμε με πραγματικά ε, μία επιπρόσθετη γραμμή ή διατρέχουμε τον κίνδυνο τους επόμενους μήνες να μάθουμε ότι η χρήση αυτών των πόρων δεν μπορεί να γίνει γιατί υπάρχει διαφορετικός προγραμματισμός και διαφορετική στοχοθέτηση έτσι ώστε να γίνουν διαφορετικές χρήσεις ή διαφορετική χρήση από την αρχικά προτιθέμενη. Δύο λεπτά για την απάντηση. Όπως σας είπα, Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε πλήρως αυτές τις δυνατότητες του κανονισμού για να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε κι εμείς. Δεν ξέρω ποια είναι η ποσοστιαία αναλογία της πολιτικής συνοχής ο πρόεδρος ε, Γιούνκερ μίλησε για 300 δις ευρώ, τα οποία θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν πλήρως. Θα πρέπει όμως να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις ιδιωτικές επενδύσεις και αναφέρθηκα στο θέμα και προγενέστερα. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν ε, τις ιδιωτικές επενδύσεις μαζί με τα δικά μας ε, κονδύλια και θα πρέπει να διαπραγματευτούμε επιχειρησιακά προγράμματα υψηλής ποιότητας έτσι ώστε να επικεντρωθούμε σε περιφέρειες που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα. Σας είπα ότι 110 δις ε, είναι η δική μας εκτίμηση για τις επενδύσεις στον τομέα της ε, καινοτομίας. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο και υπάρχουν και τα ειδικά προγράμματα καινοτομίας για τα ΕΦΗ προγράμματα και νομίζω ότι αυτά τα επιχειρησιακά προγράμματα, αν τα διαπραγματευτούμε σωστά και έχουν σαν κύριο άξονα την ανταγωνιστικότητα, για να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και επιπρόσθετες επενδύσεις, θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε τα μέγιστα για να εκπληρώσουμε τις, τους στόχους που έθεσε ο πρόεδρος Γιούνκερ. Ευχαριστώ κύριο Νίκολσον. Ευχαριστώ πολύ. Καλώ ήρθατε κυρία υποψηφία επίτροπε. Στην Βόρειο... Η Βόρειο Ιρλανδία έχει αποφεληθεί πάρα πολύ από την περιφερειακή υποστήριξη για πολλά χρόνια. Ιδιαίτερα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης υποστηρίξει την Βόρεια Ιρλανδία το 2007. Ο Επίτροπος ε, Μπαρόσο ξεκίνησε το παρόσο Task Force για να διευκολύνει την επικοινωνία με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και ε, ο στόχος ήταν να υπάρξουν περισσότερες θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη. Η Task Force ε, βρίσκεται σε μια κεντρική θέση. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι η Task Force της Ιρλανδίας θα συνεχίσει το έργο της και τη δική σας ε, θητεία. Δεύτερον, πώς βλέπετε το ρόλο της Task Force όσον αφορά την ε, ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης σε αυτή την περιοχή και τι θα κάνουν και ή θα υπάρξει μια νέα task force, η Juncker Task Force, η οποία θα μας δώσει περισσότερες δυνατότητες. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτή η Task Force για τη Βόρεια Ιρλανδία ήταν κάτι το ιδιαίτερο, ιδιαίτερα σημαντικό και συνεισέφερε για την επιτάχυνση της ειρηνευτικής διαδικασίας και της εθνικής συμφιλίωσης. Αυτή η Task Force θα συνεχίσει να υφίσταται και θα δώσει μεγαλύτερη, θα αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική γιατί θέλουμε να υπάρξει εθνική συμφιλίωση. Η Task Force θα βοηθήσει τις αρχές να δημιουργήσουν νέα προγράμματα ανάπτυξης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η σταθερότητα σε αυτή την περιοχή. Και αυτά θα πρέπει να συμβαδίσουν, δηλαδή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, οικονομική ανάπτυξη και ένα κλίμα συνεννόησης και ειρήνης, διότι όλοι μαθαίνουμε από τα διδάγματα του παρελθόντος και νομίζω ότι αυτή η Task Force για την Βόρεια Ιρλανδία, όπως και η Task Force για την ε, τουρκική, τουρκοκυπριακή και κυπριακή κοινότητα έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Θα πρέπει να υπάρξει απτή οικονομική ανάπτυξη έτσι ώστε να υπάρξει ε, παντού σωστή σύμπραξη σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Ευχαριστούμε. Η επόμενη ερώτηση είναι από την κυρία Μισελς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κρέτσου και από τη δική μου πλευρά θα ήθελα να σας καλωσορίσω θερμά εδώ στην Επιτροπή μας και θα ήθελα να αφαιρθώ στην εφαρμογή της μακροοικονομικής αρισιμότητας. Ε, τονίζετε δικαιολογημένο ότι με αυτό το εργαλείο δεν έχετε την πρόθεση να να μην ε, δώσετε τα εγκεκριμένα κονδύλια στις χώρες μέλη που είναι δικαιούχοι. Πώς θέλετε να, να αποφύγετε οι χώρες μέλη ε, στον αναπρογραμματισμό να μην ε, αγνοήσουν τα ενδιαφέροντα των Δήμων και Περιφερειών και από την άλλη πώς θέλετε να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή των Δήμων και Περιφερειών ε, στη χάραξη της περιφερειακής πολιτικής ε, τα προσεχή 7 έτη. Ή θέλετε να αφήσετε αυτή την ευθύνη στις χώρες ε, μέλη. Όπως σας είπα, η μακροοικονομική αιρεσιμότητα είναι ειπα η μακροοικονομικη ερεσιμότητα μέτρο το οποίο προβλέφθηκε την τελευταία στιγμή. Ξέρω τις ε, συζητήσεις που έγιναν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξέρω ότι πολλοί από εσάς αντιτάχθηκαν στην εφαρμογή αυτής της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας, αλλά όπως σας είπα, αυτή ήταν μια αναγκαιότητα με βάση μια κατάσταση που ζήσαμε, όπου επενδύθηκαν χρήματα χωρίς να ορίζεται το γενικό πλαίσιο. Τώρα υπάρχουν αυτές οι συνθήκες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να θεωρείται αστυνόμος ε, εναντί των κρατών μελών. Δεν είναι αυτός ο ρόλος της. Θέλει να βοηθήσει τα κράτη-μέλη, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη χωρίς την ε, πλήρωση αυτών των συνθήκων. Θα προωθήσουμε αυτό τον διαφορετικό διάλογο που προβλέπεται από τον κανονισμό. Και κάθε φορά που θα υφίσταται πρόβλημα αναστολής πληρωμών θα έρχομαι ενώπιον σας για να το συζητήσουμε. Οπωσδήποτε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. Συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας. Δεν πρέπει να πλήτεται ο πληθυσμός για κάτι που δεν πληρούν οι κυβερνήσεις, αλλά υπάρχουν πολλές προειδοποίησεις, όπως σας είπα. Δηλαδή δεν θα πει η Επιτροπή από σήμερα δεν θα έχετε πλέον χρήματα. Θα υπάρχουν προειδοποίησεις ε, ένα χρόνο πριν ή μήνες πριν, πολλούς μήνες πριν. Γιατί υπάρχουν αυτά τα χρήματα από τα ταμεία συνοχής. Έτσι κι αλλιώς διατίθενται. Σας ευχαριστώ. Και οπωσδήποτε και οι πόλεις θα πρέπει να δράσουν σε αυτό το τομέα. Ευχαριστούμε. Η επόμενη ερώτηση από την κυρία Μαντινόλφη. Ευχαριστώ. Όπως ξέρετε, πολλές χώρες της Ευρωζώνης είχαν μεγάλο προβλήματα οικονομικής διαχείρισης ε, με βάση το Σύμφωνο Σταθερότητας ως υποψήφια επίτροπος θεωρείτε ότι μπορούμε να αποκλείσουμε από το σύμφωνο σταθερότητας το ποσοστό συγχρηματοδότησης των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών και πώς θα συνεργαστείτε με τον Επίτροπο Κατάινεν. Ευχαριστώ. Γνωρίζω τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ιταλικής Προεδρίας καθώς και της Επιτροπής Περιφερειών σε σχέση με τον αποκλεισμό του συνυπολογισμού των ποσών συγχρηματοδότησης. Αυτή είναι μια απόφαση που θα ληφθεί από το Συμβούλιο. Αλλά μέχρι το Νοέμβριο πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα ευελιξίας στα πλαίσια του τρέχοντος ρυθμιστικού πλαισίου. Θα διαβιβάσω τις ανησυχίες σας στο Συμβούλιο. Χρειαζόμαστε ε, δημόσιες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που θίξατε. Δεν είναι εύκολο για ορισμένα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν ε, τη συγχρηματοδότηση μέσα στα πλαίσια των στόχων του Συμφώνου Σταθερότητας, το οποίο ενέχει περιορισμούς. Θα θέλαμε λοιπόν τα κράτη-μέλη να συνδράμουν στην χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Σίγουρα το Σύμφωνο Σταθερότητας προβλέπει κάποια ευελιξία στις δημόσιες επενδύσεις και αφήνει στα κράτη-μέλη ένα περιθώριο ελιγμών, ιδιαίτερα για τα κράτη που βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Πρόκειται για μία ε, ανησυχία γενικότερη από πολλούς εκπροσώπους κρατών μελών και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να τηρήσουμε το σύμφωνο σταθερότητας πρωτίστως, να δούμε τι δυνατότητες ευελιξίας προβλέπει και να δούμε τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο μέχρι τον Νοέμβριο σε σχέση με τον αποκλεισμό του συνυπολογισμού. Ακολουθεί η ερώτηση του κ. Στούγκερ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. μεταξύ των δέκα πιο ε, χωρών οι οποίες έχουν λάβει τα περισσότερα κονδύλια έχουν λάβει ορισμένες 8 αρνητικές κρίσεις. Τι γίνεται με τα συγκεκριμένα μέτρα. Άκουσα ως τώρα τις απαντήσεις σας και έχω αντιληφθεί ότι είστε υπέρ του διαλόγου και της συνεργασίας αλλά σκληρά μέτρα θα λάβετε. Και μπορώ να απευθύνω έκκληση προς εσάς να μας εξηγήσετε κάποιο συγκεκριμένο μέτρο, ας πούμε ένα μαύρο κατάλογο οργανώσεων ή οργανισμών που ήδη έχουν προβεί σε απάτες σε βάρος των δημοσίων χρημάτων, δηλαδή σε βάρος των επιδοτήσεων. Κάτι τέτοιο μπορεί να βοηθήσει το έργο σας. Μια μαύρη λίστα δηλαδή. Σας ευχαριστώ. Λυπάμαι. Γιατί εσείς ε, ανεβάσατε τον πύχη ως προς ε, τις απαιτήσει. Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι ιδιαίτερα δημιουργική την επόμενη περίοδο. Δεν θα επανεφεύρουμε τον τροχό. Πρόκειται για μέτρα τα οποία θα πρέπει να τηρήσουμε. Εγώ δεν μπορώ να δημιουργήσω κάτι το νέο, δεν μπορώ να δημιουργήσω νέα νομοθεσία. Εσείς ε, νομοθετήσατε και εγώ μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα τηρήσω αυτή τη νομοθεσία όπως την εγκρίνατε. Σε σχέση με το σοβαρό πρόβλημα που θίξατε, με απασχολεί το θέμα των ε, σφαλμάτων και της υπεξαίρεσης ε, δημοσίου χρήματος. Η Transparency International έχει θίξει αυτό το θέμα καθώς ε, και οι υπηρεσίες της Όλαφ. Από τις συνολικές ε, δραστηριότητες 7-13, μόνο 7% ε, σε 7% των περιπτώσεων ανέκυψαν ε, σφάλματα και πολύ μικρό ποσοστό υπεξαίρεση. Συνήθως πρόκειτο για κακοδιαχείριση, γι' αυτό θα πρέπει τα κράτη-μέλη να γνωρίζουν πώς πρέπει να διαχειριστούν τα επιχειρησιακά προγράμματα για να μην υπάρχουν σφάλματα. Από αυτή την άποψη συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί. Αλλά η Όλαφ είναι η υπεύθυνη και οι ελεγκτικές αρχές για το πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Ευχαριστώ πολύ. Ε, αναφέρεστε, αναφέρετε πολύ ξεκαθαρές ιδέες για την ε, περιφερειακή πολιτική. Ωστόσο υπάρχει ένα δημογραφικό πρόβλημα ε, που συζητά μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις. και οι, οι δημογραφικές ανισορροπίες έχουν πολύ δυσμενείς επιπτώσεις. Ε, πώς θα μπορέσουμε να επανέλθουμε στην ανάκαμψη και στην ε, εξασφάλιση θέσεων απασχόλησης. Η ολοκλήρωση της ε, περιφερειακής πολιτικής θα πρέπει να αποτελέσει εγκάρσιο στόχο ε, για όλες τις ευρωπαϊκές ε, πολιτικές. Θα πρέπει να υπάρξει μια ατζέντα για να δοθεί δημογραφική όθηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αντιμετωπίσουμε την τεράστια πρόκληση της γύρανσης ε, του, πληθυσμού και την εγκατάλειψη της υπαίθρου. Θα πρέπει η Ευρώπη να γίνει πιο ανταγωνιστική. Πώς θέλετε εσείς να συμβάλλετε στο, στην εξασφάλιση αυτού του μέλλοντος για την Ευρώπη. Uh, Φυσικά και συμμερίζομαι την άποψή σας και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση που έχει μεγάλη σημασία γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα των ε, δημογραφικών αλλαγών, της ε, απομείωσης του πληθυσμού μέχρι το 2030 ένας από τους τρεις Ευρωπαίους θα είναι άνω των 60 ετών, κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές ως προς την οικονομική μας πορεία και ανάπτυξη. Και αυτό το φαινόμενο θα μπορούσε να διευρυνθεί και από την υπογεννησιμότητα και ε, τη μετανάστευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, άλλα σημεία του πλανήτη. Άρα τα ταμεία συνοχής θα πρέπει να προετοιμάσουν το έδαφος για τα κράτη-μέλη εκεί που θα υπάρχουν προβλήματα υπογεννητικότητας. Έτσι ώστε να προετοιμάσουμε το εργατικό δυναμικό μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, καθώς και κοινωνικών υπηρεσιών, διότι όπως και νωρίτερα αυτή η κοινωνική διάσταση είναι ύψης της σημασίας. Ένα μέρος του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζει και το πρόβλημα της γύρανσης. Δεν υπάρχουν υποδομές φροντίδας και θα το δω αυτό από κοινού τον Επίτροπο Κοινωνικών Υποθέσεων για να διαχειριστούμε καλύτερα το ΕΚΤ. Ως προς το ΕΤΠΑ και τα Ταμεία Συνοχής θα πρέπει να προωθήσουμε και τις κατάλληλες υποδομές για αυτούς τους ανθρώπους. Οι δημογραφικές αλλαγές αποτελούν μείζον πρόβλημα για πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε πολύ. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον κύριο Χέτμαν. Ε, θα περάσω στην ερώτησή μου. Ε, θα δοθούν 5% του προπολογισμού στις ε, πόλεις ή προτίθεστε να, το, να αυξήσετε αυτό το όριο. Ε, θα ήθελα να επισημάνω ένα παράδοξο το οποίο προκύπτει από το Γενικό Κανονισμό 1303 που αφορά την, περιφερειακή, την ανάπτυξη πέθρου. Αυτές οι δραστηριότητες έχουν διπλασιαστεί υπό την ε, περιφερειακή πολιτική και την κοινή πολιτική γεωργίας, η οποία επίσης χρηματοδοτείται από την ε, ίδια πηγή και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο. Θα αναλάβετε κάποιες ε, δράσεις, θα κάνετε κάποιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρξει μια ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ των δύο ταμείων, ότι τα προγράμματα να μην χρηματοδοτούνται και από τις δύο αυτές πηγές. Ε, ε, γιατί αυτό ε, συνιστά πρόβλημα σε πολλές περιοχές και στην περιοχή από την οποία προέρχομαι. Έχετε δύο λεπτά για να απαντήσετε. Επαναλαμβάνω ότι οι πόλη είναι ύψης της σημασίας για την ε, περιφερειακή πολιτική και αυτό το 5% αφορά και τα κονδύλια του ΕΤΠΑ προς ολοκληρωμένα προγράμματα. Επιπροσθέτως δηλαδή από αυτά που προβλέπονται από την Γενική Περιφερειακή Πολιτική και περιλαμβάνει και πόλεις και περιφέρειες. Θα πρέπει να βρούμε τους καλύτερους τρόπους συμμετοχής των πόλεων, διότι ξέρετε ότι γίνεται αυτή η συζήτηση και πολλοί θεωρούν ότι η αρχή της επικουρικότητας είναι μία αυτόνομη αρχή. Εμείς δεν έχουμε δηλαδή κανένα δικαίωμα και δεν θέλουν νέες νομοθεσίες σε σχέση με τις πόλεις. Ενώ ε, σε άλλες περιπτώσεις ε, μας δίνουν λευκή επιταγή για τη διαχείριση. Θα πρέπει να δούμε τι θα ανακύψει από αυτή τη δημόσια διαβούλευση σε σχέση με την ε, ατζέντα των άστεων και θα ήθελα να γίνει και μία συζήτηση εδώ με βάση τις, τα συμπεράσματα από αυτή τη συζήτηση. Ως προς τη διπλή χρηματοδότηση, αυτό θα πρέπει να συζητηθεί μαζί με τον Επίτροπο για την Αγροτική Ανάπτυξη, έτσι ώστε να προβούμε σε εξοικονομήσεις και να έχουμε τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Δεν δεχόμαστε τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Thank you. Mr. Σας ευχαριστώ. Εσείς κύριε Μανσκούρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, είμαι ένας από τους τρεις εκπροσώπους ε, των υπερποντίων ε, γαλλικών εδαφών σκορπισμένη σε τρεις ωκεανούς. Άκουσα προσεκτικά την απάντησή σας σχετικά με την μακροοικονομική αρεσιμότητα. Εφιστώ ωστόσο την προσοχή σας στις καταστροφικές συνέπειες της δογματικής εφαρμογής της διατάξεως αυτής για τα υπερπόντια εδάφη, που ήδη πλήττονται από σημαντικά μειονεκτήματα που γνωρίζετε άλλωστε, και που έχουν καμιά φορά μεγάλες δυσκολίες να επιτύχουν την οικονομική ανάπτυξη στα εδάφη τους. Ερώτηση. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να επιτραπεί στα εδάφη αυτά να ξεπεράσουν τη λιτότητα και να μπορέσουν να απελευθερώσουν το αναπτυξιακό δυναμικό και κυρίως να δημιουργήσουν απασχόληση. Μπορείτε να μας βεβαιώσετε ότι θα μεταφέρετε το μήνυμα αυτό και στο μελλοντικό συλλογικό όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να ληφθεί υπόψη η πολιτική αυτή στην, στις για την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Είπα ότι συμμερίζομαι την άποψή σας και ο συνάδελφος από την ε, Ρεουνιόν μίλησε για το θέμα αυτό. Δηλαδή δεν πρέπει να πλήτεται για τις αποφάσεις που λαμβάνει η κεντρική κυβέρνηση στο Παρίσι. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το θέμα που κινούμε τον Επίτροπο Κατάινεν στα πλαίσια της οικονομικής ανάπτυξης για να βρούμε τον καλύτερο τρόπο έτσι ώστε να προχωρήσουμε. Εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους κανονισμούς που ήδη υπάρχουν. θα πρέπει να τηρήσουμε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης μέχρι ότου το Συμβούλιο αποφασίσει κάτι άλλο θα λάβουμε υπόψη την πρόταση της Ιταλικής Προεδρίας, αλλά δεν νομίζω ότι χρησιμοποιούμε το μέσο ευελιξίας που ήδη ύπάρχει στο Σύμφωνο Σταθερότητας έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των χωρών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Θα πρέπει μέσα στα πλαίσια των μακροπεριφερειών να δούμε πώς θα διατηρήσουμε τους στενούς δεσμούς με αυτές τις περιφέρειες μέσα στα πλαίσια μιας αρμονικής διαχείρισης. Και σας υπόσχομαι ότι θα προσδώσω μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα γιατί γνωρίζω ότι είναι μειονέκτημα αυτή η πολύ μεγάλη απόσταση. Πρόκειται για περιφέρειες με νησιωτικό χαρακτήρα, με γεωγραφικό έλλειμμα και μέσα στα πλαίσια του πολιετούς θα διαπραγματευτούμε ευεργετικά επιχειρησιακά προγράμματα για τις πλέον απομακρυσμένες περιφέρειες. Βεβαίως έχουν ένα, ένα ιδιαίτερο καθεστώς το οποίο έτσι κι αλλιώς σεβόμαστε. Ευχαριστώ και ακολουθεί ο κύριος Αριμό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επανέρχομαι στην αρχή της εταιρικής συνεργασίας και στην πολυεπίπεδη διακήρυση. Τα περιλαμβάνει αυτά στο άρθρο 5 ο κανονισμός και υπάρχει και κώδικας διοντολογίας ή συμπεριφορά. Για αστικά κέντρα, για ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις για να συμμετέχουν αφού πρώτα ενημερωθούν και να μπορούν να εντάσσονται έτσι τα προγράμματα. Εσείς απαντώντας γραπτός είπατε ότι θα φροντίσω να εφαρμόζεται ο κώδικας συμπεριφοράς για τις συνεργασίες. Ο καλύτερος τρόπος συνεργασίας είναι να συνεργάζονται όλα τα επίπεδα έτσι ώστε να αποφεύγονται ενδεχόμενες συγκρούσεις. Είπατε ότι η αρχή αυτή είναι ορθή εγώ συμφωνώ. Ακόμα καλύτερη θα είναι εάν εφαρμοστεί συγκεκριμένα. Και γι' αυτό έχω την εξή ερώτηση και παρακαλώ να απαντήσετε συγκεκριμένα. Πώ θα εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένα εάν η αρχή αυτή όντω εφαρμόζεται στι χώρε μέλη. Δεύτερη ερώτηση. Τι θα γίνει συγκεκριμένα εάν μια χώρα μέλο δεν σέβεται ή δεν σέβεται επαρκώς την υποχρέωσή της αυτή. Έχει κάποιο σχέδιο η δεν σεβεται επαρκω την υποχρεωση τη αυτη Επιτροπή. Thank you. We have two minutes to Δύο λεπτά απάντηση. Οι εταιρικές ε, σχέσεις υψηλής ποιότητας ε, είναι ύψης της σημασίας για τις επενδύσεις και θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή σας διότι έδωσε μεγάλη μάχη για την εισαγωγή του άρθρου 5 που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη την άποψη των τοπικών αρχών και των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα στάδια της κατάρτισης ενός προγράμματος, από τη σύλληψή του μέχρι την εφαρμογή του. Η εφαρμογή αυτού του κριτηρίου έχει μεγάλη σημασία για την κατάρτιση επιχειρησιακών σχέσεων και εταιρικών συμφωνιών. Εάν διοριστώ, από εσάς ο κύριος Χάν θα ολοκληρώσει τη διαδικασία των εταιρικών σχέσεων, αλλά τα επιχειρησιακά σχέδια θα τα προωθήσω εγώ στη συνέχεια. Και στη δική σας χώρα, στο Βέλγιο, οι συμφωνίες εταιρικές σχέσεις είναι κάτι το αυτονόητο. Υπάρχουν άλλες χώρες που δεν έχουν αυτή την κουλτούρα και ο κύριος Κοτσολίνο το έθεσε αυτό το θέμα. Δηλαδή παραπονέθηκε επειδή δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι κοινωνικοί εταίροι. Αυτό δεν ήταν υποχρεωτικό μέχρι τούδε, γι' αυτό θα παροτρύνουμε τα κράτη-μέλη στη χρήση επιχειρησιακών σχεδίων, να λαμβάνουν υπόψη τις συμφωνίες εταιρικές, εταιρικής σχέσης. Γιατί οι συζητήσεις γίνονται και σε τοπικό επίπεδο. Αυτή είναι καλύτερη εγγυήση ότι τα κονδύλια αυτά δεν θα μεταβούν σε σχέδια που δεν ανταποκρίνουν τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Δηλαδή θα, θα γίνει πληρωμή για την πληρωμή. Γιατί πολλές φορές αυτά τα σχέδια δεν ανταποκρίθηκαν στις άμεσες ανάγκες των πολιτών. Σε ορισμένες περιφέρειες χρειάζονται άμεσα επενδύσεις, χρειάζονται ε, υπηρεσίες υγείας και ούτω καθεξής. Όπως σας είπα, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων θα συνεργαστώ με μέσα στα πλαίσια τη συμμετοχής και των εταίρων. Η Επιτροπή Περιφερειών επίσης μπορεί να μας δώσει πληροφορίες γιατί εκεί υπάρχουν οι εκπρόσωποι όλων των τοπικών αρχών και πιστεύω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε την ε, συμμετοχή όλων των αρχών. Thank you. I accept the apologies, but we have to keep... Στο πολύ, συγγνώμη, ε, αλλά θα πρέπει να τηρήσουμε το χρόνο μας. Η επόμενη ερώτηση είναι από την κυρία Ρέντκε. Ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Κρέτου, αγαπητοί συνάδελφοι, οι, οι χώρες μέλη ενθαρρύνονται να συμπεριλάβουν στα επιχειρησικό τους προγράμματα περιθωριακά ποιημένες ομάδες και να φερθούν όσον αφορά τα αποτελέσματα αυτής της επένδυσης. Ιδιαίτερα η ομάδα των Ρωμά αναφέρεται στις προσωρινές διατάξει, αλλά ε, δεν είναι ξεκάθαρα κατά πόσο αυτή η ενθάρρυνση πραγματικά θα γίνει αποδεκτή από τις, αποδεκτή από τις χώρες μέλη. Πώς ε, θα εξασφαλίσει η Επιτροπή ε, ότι οι περιθωριοποιημένες ομάδες όπως είναι η Ρωμά θα συμπεριληφθούν στην πολιτική συνοχή και πώς θα διαμορφωθεί η συνεργασία με τους συναδέλφους τους ώστε να το εξασφαλίσετε. Η δεύτερη ερώτηση αφορά την αρχή μεταξύ των δύο φύλων ε, που αναφέρεται στο Γενικό Κανονισμό για, τα, για τη χρήση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το gender mainstreaming δεν περιορίζεται στο ESF, αλλά μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα ταμεία όπως είναι το Ταμείο Συνοχής. Ε, τι θα γίνει με το θέμα αυτό στο πλαίσιο της ε, πολιτικής συνοχής και πώς θα εξασφαλίσετε την ίση αντιμετώπιση των δύο φύλων. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε δύο ερωτήσεις, αλλά έχετε μόνο δύο λεπτά στη διάθεσή σας για να απαντήσετε. Um, όπως γνωρίζετε, οι ευάλωτες κατηγορίες και εκείνες που βρίσκονται στο περιθώριο θα πρέπει να μας απασχολήσουν ιδιαίτερα. Μας ενδιαφέρει η γενικότερη ανάπτυξη, αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε κανέναν πίσω. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε κάθε χρόνο, κάθε εξάμηνο μιλούσαμε για τη στρατηγική υπέρ των Ρωμά. Είναι ένα θέμα που απασχολεί ολόκληρη την Ευρώπη, δεν αφορά μόνο μερικές χώρες. Η περιφερειακή πολιτική δεν μπορεί να ασχοληθεί μόνο με ορισμένες μειονότητες ή με μία μειονότητα και τα περισσότερα χρήματα μεταβαίνουν στις λιγότερα αναπτυγμένες περιοχές, μεταφέρονται στις λιγότερα αναπτυγμένες περιοχές, εκεί που η κοινότητα των Ρωμά είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη. Εκείνοι που διαχειρίζονται τα προγράμματα πρέπει να λογοδοτήσουν στο ΕΚΤ. Γνωρίζετε ότι προέρχομαι από μία χώρα που έχει μεγάλη κοινότητα Ρωμά. Επισκέφτηκα την Ιταλία και είδα τι προσπάθειες καταβάλλονται από τις τοπικές αρχές για να αφομοιώσουν τους Ρωμά. Εκεί διατίθενται χρήματα για τους Ρωμά για να πάνε τα παιδιά στα σχολεία και είδα λεωφορεία τα οποία κάθε πρωί βρίσκονται εκεί που πρέπει και μου είπε ο αστυνόμος ε, εκεί και τότε ότι τα δικά μου παιδιά δεν έχουν λεωφορείο να τα πάει στο σχολείο, όμως τα παιδιά εδώ διαθέτουν λεωφορείο αλλά δεν θέλουν να πάνε στο σχολείο. Γι' αυτό θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες αμοιβαία έτσι ώστε να ενταχθούν αυτές οι μειονότητες. Έχουμε διαφορετικές παραδόσεις αλλά κοινού κανόνες. Τη στιγμή που τα χρήματα μίας κοινότητας ε, αφορούν μία υπηρεσία δεν θα πρέπει να ε, διασπαθίζονται αυτά τα χρήματα σε μια διαφορετική κοινότητα. Εκεί υπήρχε γενική απογοήτευση διότι αυτά τα χρήματα δεν χρησιμοποιήθηκαν σωστά. Συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Είναι ένα ε, θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε, δηλαδή να μας απασχολήσει η εκπαίδευση αυτών των κοινοτήτων Αυτή είναι και η αποστολή του Επιτρόπου Κοινωνικών Υποθέσεων, γιατί είναι μια κοινή πορεία για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ελπίζω λοιπόν να υπάρχει η βελτίωση ως προς την ισότητα των δύο φύλων. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας πω ότι Έχω δώσει μεγάλες μάχες επί του θέματος τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Χαίρομαι διότι αυτή είναι μία εξάντε αιρεσιμότητα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να τηρείται αυτός ο όρος πριν αποδοθούν τα χρήματα. Αυτό αφορά ανθρώπους με αναπηρίες και ίσες ευκαιρίες. Πρόκειται για αρχές που θα πρέπει να τηρήσουν τα κράτη-μέλη πριν τους αποδοθούν χρήματα. Και χαίρομαι διότι στα πλαίσια αυτής της αιρεσιμότητας ε, θέσατε θέματα ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε πίσω εκείνους ε, με αραπηρίες, να υπάρχει ίση πρόσβαση και των δύο φίλων και να βοηθήσουμε όλες τις μειονότητες, είτε είναι Ρωμά είτε άλλες μειονότητες. Η πρόεδρος, σας ευχαριστώ για την μακρά σας απάντηση. Ε, θα υποχρεωθώ να ε, μειώσω τον χρόνο απάντησή σας σε ένα λεπτό. Παρακαλώ λάβετε το ύψος σας. Ο κύριος Ουσπάσκιτς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα τα πω στα λιθουανικά. Ελπίζω να γίνετε επίτροπος κυρία υποψήφια διότι απαντάτε με ορθό τρόπο στις ερωτήσεις. Οι περισσότερες ερωτήσεις βέβαια είχαν ε, παρόμοιο χαρακτήρα. Μιλήσαμε για απορροφητικότητα, μιλήσαμε για προτεραιότητες των επενδύσεων. Η δική μου ερώτηση είναι λίγο διαφορετική. Θα κληθείτε να λάβετε αποφάσεις από κοινού με άλλους επιτρόπους μέσα στο συλλογικό αυτό όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ως γνωρίζετε η άμεση στήριξη επιχειρήσεων μπορεί πάντα να οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ίσως θα πρέπει να δώσουμε περισσότερα χρήματα για τη δημιουργία της ορθής υποδομής παρά να στηρίζουμε άμεσα επιχειρήσεις. Διότι έτσι θα δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο καθένας θα μπορεί να ασκήσει το επιχειρήν. Από τη δική μου εμπειρία γνωρίζω ότι τα υπόρη του προγράμματος ΣΕΠΑΝΤ οδήγησαν, οδήγησαν σε πτώχευση πολλών επιχειρήσεων. Χάσαμε τελικά περισσότερα χρήματα από όσα λάβαμε ως χρηματοδότηση. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν εδώ, έτσι ώστε τα χρήματα αυτά, οι πόροι αυτοί να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά. Παρακαλώ μόνο δύο λεπτά για την απάντησή σας. Σας ευχαριστώ, θα προσπαθήσω να είμαι, να είμαι σύντομη. Σας ευχαριστώ κύριε Ευρωβουλευτά Είμαι πεπισμένη ότι το θέμα αυτό είναι σημαντικό. Άλλωστε αυτό που θέλουμε είναι να εργαζόμαστε με αποτέλεσμα, να αποφεύγουμε τις πατάλες, περιττές πατάλες χρημάτων. Αυτό έχει σχέση βέβαια και με τις προτάσεις για τα επιχειρησιακά προγράμματα που θα υποβάλουν οι ίδιες οι χώρες μέλη. Και θα δούμε τότε εάν τα προγράμματα αυτά πηγαίνουν περισσότερο προς την κατεύθυνση της δημιουργίας υποδομών και λιγότερο προς τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Υπάρχουν βέβαια περιφέρειες στις χώρες μέλη που χρειάζονται την υποδομή, της. χρειάζονται τις υποδομές αυτές γιατί είναι στοιχείο κλειδί για την ανάπτυξή τους. Από την άλλη μεριά πρέπει να υποστηρίξουμε και τις επιχειρήσεις διότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την αληθινή ράχοκοκαλιά της κάθε εθνικής οικονομίας για τη δημιουργία απασχόλησης, για την δημιουργία ανάπτυξης. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή την κατεύθυνση, αυτό τον προσανατολισμό πρέπει να τον έχουμε πάντα υπόψη. Βεβαίως και πρέπει να στοχεύουμε σε απόδοση έργου σε σωστούς στόχους. Αλλά θα δει κάθε χώρα τι της αρμόζει καλύτερα με τις, στις ανάγκες της δηλαδή και στις ανάγκες των περιφερειών της. Πιστεύω και εγώ ότι πρέπει να επικοινωνούμε σωστά με τις χώρες αυτές μέλη, να δούμε και ποιες αλλαγές έχουν γίνει και από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι περί τα τέλη του 2015 ελπίζω, ελπίζω ότι θα μπορώ να σας υποβάλω έκθεση για την πολιτική αυτή που θα έχει στόχο συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Χέντ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα σας μιλήσω στα σουηδικά. Όπως γνωρίζετε κυρία Υποψηφία Επίτροπε, είναι πολύ σημαντικές οι διοικητικές ικανότητες της κάθε χώρας για την απορρόφηση και για τη χρήση των ταμείων. Η σωστή διοικητική ικανότητα μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή απορροφητικότητα και το χαμηλό επίπεδο των διοικητικών υπηρεσιών αντιστοίχω σε χαμηλή απορρόφηση. Πώς μπορεί να βελτιώσει κανείς την απόδοση αυτή, πώς μπορεί στο φως των παλαιότερων εμπειριών αλλά και στο φως των νέων κανονισμών, πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτή η διοικητική ικανότητα. Έχετε κάποιες ιδέες στις περιπτώσεις εκείνες δηλαδή όπου αυτό είναι αναγκαίο. Και τέλος, για την αρχή της συνεργασίας, partnership. Πώς θα την υποστηρίξετε και πώς θα υποστηρίξετε και τη συνεργασία με ιδιωτικούς οργανισμούς για να υπάρξει περιφερειακή ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτή η ικανότητα διαχείρισης είναι ακόμα μεγαλύτερες σημασίας από τα ίδια τα ταμεία και τα χρήματα που δίνουμε στα κράτη-μέλη, γιατί δεν μπορεί οι περιφέρειες και τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αυτό το πλαίσιο υπέρ των πολιτών αν ε, δεν υπάρχει σωστή διαχείριση. Η διαχειριστική ικανότητα λοιπόν έχει μεγάλη σημασία για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωστά τα κονδύλια των ε, διαφορετικών ε, ταμείων. Το θέμα αυτό είναι ύψης της σημασίας ιδιαίτερα στις περιφέρειες που δεν είναι τόσο αναπτυγμένες. και πολλές περιφέρειες δεν ήταν σε θέση να προσαρμοστούν και δεν μπόρεσαν να απορροφήσουν αυτά τα κονδύλια. Τι σημαίνει ικανότητα διαχείρισης. Σημαίνει ότι μπορεί κανείς να εφαρμόσει σωστά τους κανονισμούς έτσι ώστε τα χρήματα να φτάσουν στους δικαιούχους. Και υπήρξαν μεγάλες ε, καθυστερήσεις όπως γνωρίζετε και εσείς. Άρα ο ρόλος μας είναι να βοηθήσουμε ε, τη δημόσια διοίκηση για, ιδιαίτερα για τον έλεγχο της χρήσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θα πρέπει να υπάρχει πείρα σε αυτό το τομέα. Ίσως φαίνονται μόνο λόγια όμως, μας ενδιαφέρει η ανταλλαγή αυτή απόψεων γιατί εγώ προέρχομαι από μία χώρα η οποία βγήκε από ένα κομμουνιστικό καθεστώς και εδώ και 25 χρόνια προσπαθούμε να ανταποκριθούμε. Πολλά λειτουργούν, άλλα λιγότερο. Άρα έχει σημασία να δούμε ε, πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά αυτά τα κανονιστικά πλαίσια. Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει ε, τεχνική βοήθεια και προς τις ε, ΜΚΟ οι οποίες συνεργάζονται. Σας ευχαριστώ. Έχετε τόσα πολλά πράγματα να μας πείτε, το καταλαβαίνω, αλλά παρακαλώ τηρείτε το χρόνο σας. Ακολουθεί η κυρία Σπυράκη ευχαριστώ. Αυτή η στενότητα πιστώσεων ε, στην οποία απέληξε η οικονομική κρίση έχει μειώσει την πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Εδώ είμαι κυρία υποψηφία επίτροπε. Χρειάζονται νέα financial instruments για να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Πρώτα με την μόχλευση, με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, με την αύξηση επίσης ε, των χρημάτων που δίνονται και από την Επιτροπή. Θεωρεί η υποψηφία επίτροπος ότι τα εργαλεία αυτά πρέπει να επεκταθούν και άλλο έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες που επιβάλλει η οικονομική κρίση. Η Μελινίδα και γνωρίζετε πόσο βαριές είναι οι επιπτώσεις στις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Είμαστε άλλωστε οι πρωταθλητές της ανεργίας. Τα παραδείγματα της χρήσης των διαθωτικών ταμείων όχι μόνο για την χρηματοδότηση νέων δανείων αλλά και για την επαναχρηματοδότηση παλαιών δανείων Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστεί η υποψήφια επίτροπο στα ελληνικά. Νομίζω ότι δεν μπορώ παρά να ε, εκφράσω τη συμπαράστασή μου προς τον ελληνικό λαό, ο οποίος έζησε αυτή τη μεγάλη οικονομική κρίση και τη ζει. Η πολιτική συνοχή συνήψης της σημασίας ε, και για την Ελλάδα και για τις άλλες χώρες που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση. Οι χώρες αυτές ε, έδωσαν μεγάλο αγώνα έτσι ώστε να ανταποκριθούν σε μια κατάσταση λιτότητας και δυστυχώς έγιναν πολλές θυσίες και ως προς τις επενδύσεις. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο οι επενδύσεις είχαν αποδοτική κρίση. Χρήση, με συγχωρείτε, γνωρίζω ότι το 70% των ε, επενδύσεων στην Ελλάδα αφορούν τον δημόσιο τομέα. Όμως ε, θα πρέπει να δούμε το σημαντικό ρόλο των χρηματοδοτικών μέσων έτσι ώστε ιδιαίτερα για τις νέες γενναίες να προσδώσουμε την κατάλληλη σημασία ως προς τη χρήση αυτών των επενδύσεων και να υπάρχει και περιθώριο ελιγμών και για επιπρόσθετες επενδύσεις, ιδιαίτερα στους δύσκολους αυτούς καιρούς όπου το δημόσιο χρήμα είναι περιορισμένο. Σίγουρα θα πρέπει να ε, υπάρξουν υπηρεσίες ε, αρρωγής και φυσικά η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να μας απασχολεί ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ. Τανκίλα. Πιστεύω σε σένα Κορίνα και πιστεύω ότι γνωρίζεις πολύ καλά τις αρχές συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Ως Επίτροπος για Περιφερειακά Ζητήματα και Ανάπτυξη είμαι σίγουρη ότι θα προσδώσεις μεγάλη σημασία στην ε, ε, διόρθωση των σφαλμάτων ιδιαίτερα. Τι προβλέπετε για την μείωση των σφαλμάτων στα επιχειρησιακά προβλήματα και επιχειρησιακά προγράμματα, με συγχωρείτε, για την περίοδο 2007-2014. Πώς θα επανορθωθούν αυτά τα ασφάλματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ευγενικά σου λόγια. Όπως είπα, τα σφάλματα αυτά αποτελούν το 7% των συνολικών προγραμμάτων την περίοδο 7-14 και αφορούν τις επενδύσεις των διαρθρωτικών ταμείων ιδιαίτερα. Θα πρέπει να εγκρίνουμε μέτρα για να μειώσουμε το ποσοστό σφαλμάτων. Από το 7% μόνο το 1% αφορούσε απάτες οι οποίες ε, τώρα εξετάζονται. Όσον αφορά την απάτη, τα μέτρα είναι σαφή. Γίνεται ανάκληση επενδύσεων, αναστολή και ανάκληση όταν αποδειχτεί η απάτη. θα πρέπει να αποδώσουμε λογαριασμό στον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Γι' αυτό και φέρουμε την ευθύνη να επαγρυπνήσουμε ως προς την χρήση αυτών των χρημάτων. Από την άλλη πλευρά, τα περισσότερα λάθη είναι διοικητικά ασφάλματα από άγνοια του κανονισμού, μη σωστή εφαρμογή του και όπως σας είπα θα πρέπει πρέπει άμεσα να ασχοληθούμε με αυτά τα ζητήματα. Στη δική μας περιφέρεια υπήρξαν προβλήματα ως προς τις δημόσιες προμήθειες και η Επιτροπή θα αποστείλει οικονομολόγους επιτόπου για να βοηθήσουν τους εθνικούς εμπειρογνώμονες εκεί που χρειάζεται βοήθεια, δηλαδή για αποφυγή σφαλμάτων. Θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, αλλά φυσικά δεν αποκλείουμε τις περιφέρειες και τα κράτη-μέλη στην απόδοση. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μπόγκοβιτς, παρακαλώ. Κυρία υποψήφια επίτροπε, έρχεσαι από τη Ρουμανία, εγώ είμαι από τη Σλοβενία και πιστεύω ότι και οι δύο χώρες είναι γνωστές για τις δυσκολίες που έχουν να πάρουν ευρωπαϊκά κονδύλια. Γι' αυτό έχουμε την εντύπωση ότι η δυνατότητα απορρόφησης εκ μέρους των ευρωπαϊκών χωρών είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Αναφέρατε ορισμένα εμπόδια τα οποία θα πρέπει να καταργηθούν, για παράδειγμα, κατά την προετοιμασία προγραμμάτων κλπ. Νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε προγράμματα εταιρικής ε, συνεργασίας, ε, ε, επιχειρησιακά προγράμματα κλπ εσείς ως Επίτροπος έχετε μία ενεργητική προσέγγιση. Νομίζω δεν θα πρέπει να υπάρχουν ασυνέχειες και καθυστερήσεις στις πληρωμές. Η Επιτροπή βεβαίως θα πρέπει να παράσχει τη δική της συνδρομή, αλλά θα πρέπει να ασκεί και πίεση στις χώρες ε, μέλη για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Ε, τι κάνετε από την έννοια αυτή. Ευχαριστώ. Φυσικά τα τελευταία χρόνια τα κράτη, ορισμένα κράτη-μέλη αντιμετώπισαν προβλήματα. Όμως έχουν υπάρξει βελτιώσεις. Εμείς έχουμε εγκρίνει κανονισμούς που θα τεθούν σε εφαρμογή. Τα κράτη-μέλη όμως ε, πρέπει να είναι πολύ πιο ευσυνείδη τα τα κράτη-μέλη πρέπει ε, να αποδώσουν λογαριασμό. Δεν θα πρέπει όμως όλα να τα θυσιάσουμε στο βωμό της ταχύτητας και της ταχείας εφαρμογής. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και να απορροφηθούν σωστά αυτά τα κονδύλια θα πρέπει να μην υπάρχει κατακαιρματισμός των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας, ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια του ΕΤΠΑ. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι θα βασιστούμε στις επενδύσεις ε, για την καινοτομία, στην ψηφιακή ατζέντα, στις ΜΜΕ και στην οικονομία μειωμένων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Υπάρχουν πολλές αιρεσιμότητες που θα βοηθήσουν τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα των ε, ευρωπαϊκών κονδυλίων. Δεν θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της διοικητικής ικανότητας, διότι αναφέρθηκα ήδη. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό και από τα χρήματα τα ίδια, διότι τα χρήματα αυτά δεν απορροφήθηκαν. Υπάρχουν διαρθρωτικές ελλείψεις. Εγώ είμαι αισιόδοξη παρόλα αυτά και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να οθήσουμε τα κράτη-μέλη έτσι ώστε μέχρι το τέλος του 2015 να αποπληρώσουν τα, τα δάνεια αυτά. ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υποψήφια Επιτροπέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποσχέθηκε να υποστηρίξει την Ουκρανία. Αυτό δεν θα προσφέρει τίποτε όμως αν εξακολουθήσει το ε, οδικό δίκτυο της Ουκρανίας να είναι αποσυνδεμένο από το ευρωπαϊκό. Δεν υπάρχουν απαραίτητοι διάδρομοι μεταξύ Ουκρανίας και Ανατολικής Ευρώπης που θα έπρεπε να περνά από την Πολωνία και από τις ανατολικές της περιφέρειες όπως το Λούμπλιν που εκπροσωπώ εγώ εδώ. Η ερώτησή μου έχει ως εξής. Κυρία Υποψηφία Επίτροπε, θα υποστηρίξετε δράσεις εντός της ε, πολιτικής συνοχής για επενδύσεις και για τη δημιουργία του ε40 και των υδάτινων οδών. Παρακαλώ να είναι σύντομη η απάντησή σας. Ευχαριστώ βεβαίως. Όλοι είμαστε αλληλέγγυοι προς τον Ουκρανικό λαό η χώρα αυτή προσβλέπει στην προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς ε, ελήφθη αυτή η απόφαση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής να μην διευρύνει το πολιτικό χώρο για τα επόμενα πέντε χρόνια. Εμείς φέρουμε μεγάλη ευθύνη, έχουμε προγράμματα τα οποία αφορούν αυτές τις περιφέρειες, γιατί πρόκειται για μακροπεριφέρειες, πρόκειται για περιφέρειες στο, στα πλαίσια της ε, διαδικασίας σύνδεσης και πριν από την ένταξη θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις ανάγκες είτε πρόκειται για τη Σερβία για τη δημοκρατία της Μολδαβίας ή την Ουκρανία. Στα πλαίσια της στρατηγικής ε, του Δούναβη εντάσσεται και η Ουκρανία. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε συγκεκριμένη δράση για να υποστηρίξουμε τον πληθυσμό αυτής της περιοχής. Ε, παράλληλα, τα προγράμματα υποδομής είναι ύψης της σημασίας. Ξέρετε ότι ένα μεγάλο μέρος των κονδυλίων συνοχής σχετίζονται με τις ε, υποδομές. Θα το συζητήσω και με τον Επίτροπο Χάν που ασχολείται με την πολιτική γειτονία και με την Γενική Διεύθυνση Μεταφορών για να έχουμε μια συνολική εικόνα και να δούμε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη τα κατάλληλα μεταφορικά μέσα και προώθηση των υποδομών στον τομέα των μεταφορών. Και για τις Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Η κυρία Βαλίνα παρακαλώ. Sorry. Bien, buenos días, señora. Καλημέρα σας, ε, κυρία Κρέντο. Ε, αναμφίβολα υπάρχουν πολλές ε, κοινότητες που πάσχουν από καθυστερήσεις στις ε, πληρωμές, ε, στις υποχρεώσεις πληρωμών. Και από την άλλη υπάρχουν οι νέες διατάξεις, κοινές διατάξεις, το άρθρο 23, όπου εξαγγέλλεται η μακροαιρεσιμότητα των κονδυλίων και οι περιφέρειες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια αν δεν εκπληρώνουν ε, τους όρους, κάτι που είναι αδύνατο για μας, γιατί ε, οι κοινότητες λαμβάνουν μόνο το 10% του προϋπολογισμού. Ε, και έχουν γίνει περικοπές και είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως σας είπα, να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στα διαρθωτικά ταμεία. Uh, uh, Έχω απαντήσει στην πρώτη ερώτηση του κυρίου Βανίστελ Ρόι ως προς το χάσμα αυτό ε, στις πληρωμές Έχουμε 23,4 δις που δεν έχουν καταβληθεί λόγω μη απορρόφησης και γίνεται μια σοβαρή συζήτηση για τον ε, τρόπο εξέβρεσης ε, μιας ε, λύσης για να αποφύγουμε αυτή την καθυστέρηση πληρωμών και την ε, καθυστέρηση της εφαρμογής των ε, επιχειρησιακών προγραμμάτων. Είναι προβλήματα που έχουν ανακύψει εξαιτίας της καθυστέρησης ε, πληρωμών. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε και την δική σας υποστήριξη μέσα στα πλαίσια του διορθωτικού προϋπολογισμού για το 2015 για να αποφύγουμε ε, τη μία απορρόφηση ως προς την μακροαιρεσιμότητα, όπως σας είπα, το Συμβούλιο και η Επιτροπή αποφάσισαν. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να προβλέψω την αναλογική εφαρμογή και την ίση μεταχείριση μεταξύ κρατών μελών. Εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή θα μπορέσει να συμμετάσχει στις συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τις ενδεχόμενες αναστολές. Ελπίζω σε καμία περίπτωση να μην φτάσουμε σε αυτή τη δυσχερή στιγμή αλλά θα σας δώσουμε όλες τις πληροφορίες πριν από την αναστολή πληρωμών. Αυτή η μακροοικονομική ρήτρα διασφάλισης είναι ε, η τελευταία, ε, το τελευταίο βήμα στο οποίο θα καταφύγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την τήρηση της μακροαιρεσιμότητας. Grazie. Concordo con i miei σύμφωνο. ως προς το θέμα της αντιμετώπισης της απάτης και ελπίζω να ληφθούν έγκαιρα μέτρα για να μπορέσουμε αποδοτικά να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Θα ήθελα να σας μιλήσω όμως για τις αξιολογήσεις των παρεμβάσεων του παρελθόντος στα πλαίσια της πολιτικής σύνοχης. Πρόκειται για ποσονικά μέτρα, δηλαδή τη δυνατότητα δαπάνης των κονδυλίων ανάλογα με τα έργα που έχουν επιτελεστεί. Πώς θα διαρθρώσετε το νέο σύστημα αξιολόγησης για τη νέα περίοδο προγραμματισμού. Κρέτσου. Καταρχήν αναφερθήκατε στη διαφάνεια. Καθίσατε σαφές ότι θα πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή έναντι της απάτης. Θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ Γενικής Δεύθυνσης Ρέτζιο και Όλαφ ε, έτσι ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Δηλαδή και, μέτρα, και προληπτικά μέτρα και διορθωτικά μέτρα. Ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση της απάτης και θα, θα χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες της Transparency International μέσα στα πλαίσια των δημοσίων προμηθειών ιδιαίτερα. Θα υπάρξει και τεχνική αρρωγή για την ε, σωστή χρήση των πόρων. Και όπως είπατε θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό ως προς τις αξιολογήσεις. Για μένα το πιο σημαντικό κριτηρίο είναι η προστιθέμενη αξία αυτών των προγραμμάτων σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Είναι το πιο σημαντικό κριτήριο το οποίο ε, χρειαζόμαστε σε αυτή την περίοδο της κρίσης. Δεν θα θυσίαζα ποτέ την ποιότητα βεβαίως για να έχουμε καλύτερη απορροφητικότητα για να αυξηθεί ο δείκτης απορροφητικότητας. Θα πρέπει να υπάρχει πραγματικά προστιθέμενη αξία. Και όπως σας είπα, μας ενδιαφέρει και το θέμα της χρήσης του δίκτυου του web. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που με ενδιαφέρει είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με βάση τα προγράμματα αυτά. Ευχαριστώ. Η επόμενη ερώτηση, η ερώτηση του κυρίου Παπαδάκη. Κρέτσου, στη χώρα μου την Ελλάδα, τα πάνω από 20 δις της περίοδου 2007-2013 δόθηκαν για την κατασκευή υποδομών και έργων που έχουν ανάγκη επιχειρηματική όμιλη και η κερδοφορία τους. Ενώ απορρίφθηκαν ως μη επιλέξιμα για τις λαϊκές ανάγκες έργα όπως αντιπλημμυρικά, αντισυσμικά προγράμματα, προγράμματα κατασκευής λαϊκής στέγης, σχολείων και νοσοκομείων. Με το λαό να ζει μέσα στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Επιπλέον με τον εκβιαστικό όρο περί στο εξή τα κονδύλια θα διακόπτονται αν ένα κράτος μέλος δεν ακολουθεί τα αντιλαϊκά μέτρα που προβλέπονται με το ευρωπαϊκό εξάμενο και με την ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση. Πώς τοποθετήστε στη χρησιμοποίηση των κονδυλίων ως εργαλείο για την επιβολή βάρβαρων αντιλαϊκών μέτρων που προβλέπονται από τα μνημόνια διαρκείας που σχεδιάζουν από κοινού Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσει για όλα τα κράτη-μέλη της. Ευχαριστώ. I would like to ask you for a very short answer. Να συζητήσω να είστε πολύ σύντομοι. Επαναλαμβάνω ότι όταν μιλάμε για τις μακροπεριφέρειες και τη μακροαιρεσιμότητα, μιλάμε για έκτακτες συνθήκες. Σας υπόσχομαι ότι θα επανέλθω να συζητήσουμε μέσα στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου όταν ανακύψει ανάγκη. Ως προς τις φυσικές καταστροφές, εδώ κινούμαστε στα πλαίσια του, των Ταμείων Αλληλεγγύης για την διαχείριση καταστάσεων κρίσης. Αντιμετωπίσαμε παράλληλες και παρόμοιες περιστάσεις στη δική μου περιφέρεια και σίγουρα όταν πλήττεται ο πληθυσμός θα πρέπει να ανακουφίζεται. Είμαι αλληλέγγυα με τις μεσογειακές οικονομίες, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ελλάδα που επλήγησαν και νομίζω ότι η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής οδήγησε σε καταπράνηση κάπως της κατάστασης. Ελπίζω αυτό να έχει συνεχιστεί. Και κατανοώ ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να ανταποκριθούμε και μέσα στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας, αλλά το Σύμφωνο Σταθερότητας παρέχει ένα περιθώριο ελιγμών και είμαι και εγώ πολύ περίεργη να δω, όπως και εσείς, τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο Υπουργών του Νοεμβρίου. Η κυρία Σμόλκοβα. Mám identickú otázku, ako už povedal môj kolega z Polska v úvode, takže nebudem ju... Ναι, δεν πρόκειται να επαναλάβω την ερώτηση του συναδέλφου από την Πολωνία. Η δική μου ερώτηση αφορά τη στρατηγική για τα Καρπάθια. Για μας, ε, ερχόμαστε από την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία ασφαλώς, αυτή η στρατηγική είναι εξαιρετικά σημαντική. Ε, ε αυτή τη στιγμή οι χώρες αυτές συνεργάζονται συχνά σε πολλούς ε, τομείς. Ευχαριστούμε, λοιπόν περισσότερες πρωτοβουλίες από τις χώρες μέλη, όχι να αρχίσουν από την αρχή. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν ε, πολλές ε, πρωτοβουλίες και οι Ευρωπαϊκές μπορούν να μας στηρίξουν. Έχετε την πρόθεση να επισκεφτείτε συγκεκριμένες περιφέρειες για να δείτε πώς εκταμιεύονται τα κονδύλια και πώς απορροφούνται. Ε, θα μπορούσατε να έρθετε στην ε, Σλοβάκια, την Πολωνία, την Ουγγαρία και την Ουκρανία ε, και θα δείτε πώς μπορεί η στρατηγική των Καρπαθίων να μας βοηθήσει οι στρατηγικές, οι μακροπεριφερειακές είναι βιώσιμες διότι κινητοποιούνται όλα τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν για να ξεπεράσουν τις προκλήσεις της κάθε περιφέρειας. Αλλά η πρωτοβουλία θα πρέπει να προέρχεται από τα κράτη-μέλη από το υψηλότερο δυνατό επίπεδο η στρατηγική του Δούναβη προήλθε από μία επιστολή του Πρωθυπουργού της Ρουμανίας και της Αυστρίας. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να συζητήσουν αυτές τις στρατηγικές, τη στρατηγική των Καρπαθίων μεταξύ άλλων. Θα πρέπει να κινητοποιήσουμε τις εμπλεκόμενες περιφέρειες και τις τοπικές αρχές αυτών των περιφερειών, διότι οι τοπικές αρχές γνωρίζουν πολύ καλά πώς μπορούν να ανταποκρινθούν στις ανάγκες. Δεν νομίζω ότι εμείς από Βρυξέλλες ξέρουμε τι συμβαίνει στη Φλοβακία ή τι συμβαίνει στη Βαλτική ή στα, στην Ιόνιο, στο Ιόνιο Πέλαγος. Θα, θα πρέπει να προέλθουν οι πρωτοβουλίες από τα κράτη-μέλη. Ως προς την πρόσκλησή σας, προτίθεμαι να επισκεφθώ το μεγαλύτερο μέρος των 277 περιφερειών που υπάρχουν. Η κυρία Ντανούτα Χούμπνερ κατάφερε να επισκεφθεί όλες τις περιφέρειες και τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν λίγο μικρότερη. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα θα επισκεφθώ τις περιφέρειες ε, που είναι οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι αυτών των κονδυλίων και που τα χρησιμοποίησαν με επιτυχία. Αλλά θα ασχοληθώ και με τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες γιατί έχουν ε, τις μεγαλύτερες ανάγκες θα μεταβώ και εκεί με τους διευθυντές της Γενικής Διεύθυνσης Ρέγγιο. Δεν θέλω να υπάρξουν κυρώσεις, θέλω να βοηθήσουμε, γιατί αυτό περιμένουν οι άνθρωποι από εμάς, οι πολίτες από εμάς. Να υπάρχει σωστή χρήση αυτών των χρημάτων. It Ήταν πολύ σημαντικό ε, που σας ακούσαμε, αλλά έχουμε μια καθυστέρηση 25 λεπτών και θα ήθελα να παρακαλέσω τους επόμενους 10 ομιλητές που θα υποβάλουν ερωτήσεις, παρακαλώ να είναι πολύ σύντομοι. Ε, και για τις απαντήσεις, ε, κυρία Επίτροπε, θα σας δώσω ένα λεπτό. Η επόμενη ερώτηση είναι από την κυρία Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ε, πολλές επιφυλάξεις όσον αφορά τις ε, γραφειοκρατικές και διοικητικές ε, διαδικασίες που συνδέονται με την χορήγηση των κονδυλίων. Το, οι έρευνες του Euro, οι δημοσκοπήσεις του Eurobarometer λένε ότι έχει μειωθεί η αξιοπιστία των Ευρωπαίων πολιτών. 50% θεωρούν ότι η διαφθορά είναι σημαντικό πρόβλημα και οι στατικές της Όλαφ του 2013 λένε ότι οι εκθέσεις για την ε, διαφθορά στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων αυξάνονται συνεχώς. Μια και έγινε επανελειμμένα μνήμα στη δαφάνεια, παρακαλώ να μου απαντήσετε συγκεκριμένα ε, ποια, πώς θα διαμορφωθεί συγκεκριμένη συνεργασία με την Όλαφ και ποια είναι τα σχέδια της Κομισιόν όσον αφορά την ε, δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελία και πώς ε, βλέπετε το ρόλο των ε, πολιτών σε πρωτοβουλίες κατά πολέμησης της διαφθοράς και της απάτης. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η σωστή χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων αφορά την δική μας ευθύνη δεν μπορούμε να χάσουμε την αξιοπιστία μας ή την εμπιστοσύνη των πολιτών εξαιτία αυτών των περιπτώσεων που δεν μπορούν να γίνουν δεκτές. Η Ρέγγιο συνεργάζεται στενά με την Όλαφ για την καταπολέμηση της απάτης και θα λάβουμε μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας σε περιπτώσεις όπου διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ελλείψεις. Αλλά ελλείψεις δεν σημαίνουν απάτη. Έχει μεγάλη σημασία η εμπιστοσύνη των λαών, η οποία δεν εξαρτάται μόνο από την περιφερειακή πολιτική. δημιουργήσαμε δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, αλλά υπάρχουν και ε, εκατοντάδες ε, χιλιάδες επιχειρήσεις που άρχισαν τη δραστηριότητά τους, έκαναν έναρξη δραστηριότητας εξαιτίας, ε, μάλλον χάριν στα κονδύλια που εμείς έχουμε αποδώσει. Κύριε <clears throat> Σώσα Βάγνερ, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Υποψηφία Επίτροπε, ε, πολύ συνοπτικά θα σας υποβάλω την ερώτησή μου. Τα διευθυντικά ταμεία και όλα τα άλλα ταμεία της Ευρώπης ε, ε, ε, προβλέπουν πάρα πολλά κονδύλια για τους πολίτες. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη από μέρους σας ούτως ώστε οι πολίτες να είναι βέβαιοι ότι αυτή είναι μια μορφή δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Γιατί, και ότι η απασχόληση δημιουργείται ε, ακριβώς μέσω της, απασχόλησης, μέσω της ε, χρησιμοποίησης αυτών των κονδυλίων. Δεύτερον, τι σκέφτεστε εν σχέση με την θολή ερμηνεία όσον αφορά τις αρχές διαχείρισης και τις αρχές ελέγχου. Εδώ υπάρχει μία σύγχυση και τα άτομα τα οποία ενέχονται στην, ε, τα οποία ε, εργάζονται στο πλαίσιο των ταμείων καταγγέλουν ακριβώς αυτή τη σύγχυση. Συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε την επικοινωνία με βάση τους κανονισμούς που διαθέτουμε. Υπάρχουν περιφέρειες που δεν γνωρίζουν τους πλέον διαφανείς κανόνες που ισχύουν τώρα για την απορρόφηση των πόρων και δεν κοινοποιήσαμε αρκετά τα ευεργετήματα της πολιτικής συνοχής. Αυτά τα απτά αποτελέσματα δηλαδή της ε, πολιτικής συνοχής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν 594.000 θέσεις εργασίας, 77.000 επιχειρήσεις άνοιξαν τη δραστηριότητά τους, ε, δημιουργήθηκαν νέες οδικές και σιδηροδρομικές αρτηρίες, 25.800 ε, χιλιόμετρα και πρόσβαση στους υδάτινους πόρους, καθώς και ευρυζωνικά δίκτυα για 8 εκατομμύρια κατοίκους. Θα πρέπει λοιπόν να υπενθυμίζουμε αυτά τα αριθμητικά στοιχεία για να κατανοήσουν οι πολίτες πώς έχουν ευεργετηθεί. Το 85% αυτών των προγραμμάτων χρηματοδοτήθηκαν από εμάς, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εσείς κύριε Ποστινάρο. Η εξοικονόμηση της ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση είναι ο καλύτερος ε, τρόπος διασφάλισης της ενεργειακής αυτονομίας, ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια των σχέσεων με τη Ρωσία και του επαναπροσδιορισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση της ε, στρατηγικής ενέργειας. Επειδή το ΕΤΠΑ και τα Ταμεία Συνοχής έχουν ε, προωθήσει το θέμα της επιλεξιμότητας των σχεδίων για τις ανανεώσιμες και την ε, ενεργειακή αποδοτικότητα, τι προτίθεσαι να κάνεις για τις περιφέρειες και για τις δικές μας ε, περιφέρειες, για την ευφύ χρήση των κονδυλίων έτσι ώστε το κοινωνικό πακέτο να διασφαλίσει την ενεργειακή, να προωθήσει την ενεργειακή ασφάλεια. Θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή σας διότι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ε, προώθηση πολιτικής συνοχής και της ε, ενέργειας. Ξέρετε ότι προωθούμε την ενεργειακή αποδοτικότητα και αυτονομία μας. 38 ε, δις ευρώ έχουν αποδοθεί για την ενεργειακή απόδοση και τη μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε σχέση με τη στέγη και την ε, και ανανεώσιμες. Στην παρούσα γεωστρατηγική συγκυρία θα πρέπει να επενδύσουμε στις ανανεώσιμες και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε βεβαίως και σε θέματα ενεργειακής ασφάλειας. Thank you. And the next question, Mr. Zeller. Ευχαριστώ πολύ. Την επόμενη ερώτηση θα αποβάλει ο κύριος Τσέλερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κρέτσου. Ένα από τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι τα σύνορα για τους ε, πολίτες δεν γίνονται πλέον αισθητά, μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Αλλά εκεί όπου θέλουν να συνεργαστούν με μεθοριακές ε, ε, περιοχές ε, βλέπουμε ότι οι πόλεις τις εμποδίζουν σε αυτό. Και φτιάξαμε ένα νομικό εργαλείο το οποίο έχει διευρυνθεί στην προηγούμενη θητεία, την Ευρωπαϊκή Ένωση για Εδαφική Συνεργασία. Εσείς ε, πρόκειται να προσπαθήσετε αυτό το εργαλείο να γίνει το καθοριστικό εργαλείο ε, συνεργασίας ε, και εκεί όπου τα εθνικά κράτη ε, παρεμποδίζουν ε, την περιφερική αυτή συνεργασία να εξαλείψατε αυτές τις αντιστάσεις, τις αντιδράσεις. Ο κύριος Χάν γνωρίζει αυτό το μέγεθος και θα σας συνδράμει. Τα επόμενα δύο χρόνια θα πρέπει να παλέψουμε ούτως ώστε η πολιτική συνοχή να έχει ένα μέλλον. Στην αρχή της ε, προηγούμενης θητείας έμοιαζε να θέλουμε να, να, να, να θυσιάζεται η, η πολιτική συνοχή χάρη της περιφερειακής πολιτικής. Εσείς ε, θα φροντίσετε ούτως ώστε η πολιτική συνοχή να έχει ένα βιώσιμο μέλλον και μετά το 2020. Σας ευχαριστώ. Μπορούμε να διαβούμε τα σύνορα, όπως ξέρουμε, αλλά υπάρχουν διαφορετικοί αναπτυξιακοί ρυθμοί. Πιστεύω ότι αυτά τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας δημιουργήθηκαν για να θεραπεύσουν και είδα πολύ ωραία παραδείγματα. Ιδιαίτερα μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας οικοδομήθηκε ένα νοσοκομείο. Το ίδιο αφορά στα σύνορα Ρουμανίας και Ουγγαρίας. Εσείς όμως αναφερθήκατε και στην εδαφική ολοκλήρωση, την κοινή βοήθεια. Πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αφήσουν τις τοπικές αρχές να δράσουν και να μην υπάρχει τόσο ισχυρός παρεμβατισμός προς τις περιφέρειες, διότι οι περιφέρειες γνωρίζουν ε, καλύτερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ως προς το μέλλον της ε, πολιτικής ε, συνοχής, θα ήθελα να σας πω ότι γνωρίζω όλες τις επιθέσεις που δέχεται η πολιτική συνοχής. Πολλοί επιθυμούν να μειωθούν τα κονδύλια. Εμείς θεωρούμε ότι μέχρι το 2020 πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η περιοχή για την εξάλληψη των ανισορροπιών. Όλοι έχουν να κερδίσουν από αυτό. Θα ακολουθήσει η ερώτηση του κυρίου Ροπέ. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, κυρία Υποψήφια Επίτροπε. Αρχίζουν και παραλαμβάνονται βέβαια οι ερωτήσεις σε κάποιο βαθμό. Συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι η χρηστή διαχείριση είναι προϋπόθεση για την ορθή εφαρμογή πολλών πολιτικών. Όπως προκύπτει από την πράξη, τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν συμμετέχουν οι περιφερειακές αρχές σε διάφορες εταιρικές σχέσεις ποιο ρόλο θα παίξετε έτσι ώστε να βελτιώσετε την περιφερειακή διαχείριση και ποια μέτρα θα λάβετε για να επιτύχετε την αποκέντρωση στην πράξη. Μπορείτε να παριθμίσετε ορισμένα συγκεκριμένα μέτρα που προτίθεστε να λάβετε. Η καλοδιαχείριση είναι ύψης της σημασίας για τα ταμεία συνοχής. Ε, η συμμετοχή των τοπικών αρχών αποτελεί απαράβατο όρο για τη συμμετοχή τους. Σίγουρα θα γίνει μία μελέτη για να δούμε πώς θα εφαρμοστεί η εταιρική σχέση. Υπάρχει ένας κώδικας συμπεριφοράς Υπάρχουν περιπτώσεις και περιπτώσεις, υπάρχουν χώρες που έχουν αποκεντρωθεί και άλλες όχι. Άλλες χώρες καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για αποκέντρωση. Θα πρέπει το θέμα να συζητηθεί με κάθε κράτος ε, ξεχωριστά, γιατί υπάρχουν διάφορα επίπεδα ανάπτυξης. Ακολουθεί η ερώτηση του κύριου Νίκολσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτόπου, στην πράξη, πολλοί έχουν εκφράσει και προς εμένα ανησυχίες για υλοποίηση έργων επιτόπου. Έχουν εκφράσει ανησυχίες για τις αρνητικές επιπτώσεις νέων προγραμμάτων που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια τεχνογνωσίας. Είναι λοιπόν σημαντικό να μην χαθούν οι, ε, τα μέχρι τώρα επιτεύγματα από ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην υλοποίηση νέων έργων. Τι θα κάνετε για να εξασφαλίσετε μια ομαλή μετάβαση έτσι ώστε τα ταμεία να αρχίσουν να έχουν θετικές συνέπειες στις ενδιαφερόμενες κοινότητες όσο το δυνατόν ταχύτερα και έτσι ώστε να βασιστούν και στα παλαιότερα επιτεύγματα. Ευχαριστώ. Υπάρχει αυτή η νέα διάρθρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ορίστηκε από τον πρόεδρο Γιούνκερ, όπου θα συνεργαστούμε με όλους τους υπεύθυνους ε, για τα διαφορετικά ταμεία και τα επενδυτικά. Η Γενική Διένθηση Ρέγγιο είναι υπεύθυνη για τα περιφερειακά ταμεία και το, τα Ταμεία Συνοχής και θα συνεργαστούμε με τον Επίτροπο Κατάινεν για να φτάσουμε στα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. Έχει μεγάλη σημασία να προωθήσουμε τα επιχειρησιακά προγράμματα για την περίοδο 14-20. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το μέλλον για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτά τα προγράμματα. Θα πρέπει βεβαίως να κλείσει με επιτυχία η περίοδος 7-13 γιατί ξέρετε ότι υπολείπονται πληρωμές. Θα πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε με τη νέα αυτή περίοδο προγραμματισμού. Thank you. Η Σας ευχαριστώ. Ακολουθεί η ερώτηση του κυρίου Αμπαούνθ. Καλημέρα σας, κυρία Κρέτου. Θα ήθελα να επιμείνω εδώ βρίσκομαι. Θα ήθελα να, επι... Ε, να επιμείνω στο θέμα της διασυνορικής συνεργασίας. Ε, εσείς θέλετε να την ενισχύσετε, αλλά δεν νομίζω ότι ο προϋπολογισμός θα ε, σας βοηθήσει. Ε, στην περίπτωση της χώρας των Βάσκων, θα πρέπει να γίνουν πολλές προσπάθειες ε, για να ξεπαραστούν ε, τα εμπόδια. Και νομίζω ότι η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει να είναι το πιο σημαντικό κομμάτι αυτής της ε, συνεργασίας. Στην Ιρλανδία, όπως και στην Ιρλανδία, στη δική μου χώρα τα ευρωπαϊκά διασυνοριακά προγράμματα θα πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη σταθερότητα και την ειρήνευση και την επίλυση της σύγκρουσης. Εσείς γνωρίσατε, αναγνωρίσατε αυτό το ρόλο και ε, επίσης υπάρχει και Κύπρος. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμοστεί ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ε, τι θα κάνετε για να προωθήσετε λοιπόν την διαπεριφερειακή ε, συνεργασία και τη διασυνοριακή συνεργασία. Με, μεγάλα, με μεγάλη χαρά θα επισκεφθώ την χώρα των Βάσκων για να δω άμεσα ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Το ζήτημα αυτό θα πρέπει να το δούμε και με τις αντίστοιχες περιφέρειες και με την κεντρική για να υπάρχει κοινή κατανόηση μεταξύ περιφερειών και κυβέρνησης. Υπάρχουν περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο. Γι' αυτό μιλώ για τις πληγές της ιστορίας. Εμείς μέσω της πολιτικής συνοχής μπορούμε να ε, οδηγήσουμε τους, τους ανθρώπους στο να συμφιλιωθούν. Τώρα συνεργάζεστε για την οικονομική ανάπτυξη και για την απασχόληση. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεπεράσει κανείς τις πληγές του παρελθόντος που πολλοί έχουμε ζήσει. Η διασυνοριακή συνεργασία έχει μεγάλη σημασία. Πολλά μπορεί να γίνουν και από τις δύο πλευρές των συνόρων και σας ε, έδωσα παραδείγματα, αυτά παραδείγματα. Έθεριτς, θα προσπαθήσω να βοηθήσω, θα κάνω μια ερώτηση που μπορείτε να την απαντήσετε πολύ γρήγορα. Ελπίζω να πείτε ναι. Προέρχομαι από τα West Midlands στο Ενωμένο Βασίλειο που όπως λέει και το BBC έχουν περισσότερη φτώχεια από οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια του Ενωμένου Βασιλείου. 21% του πληθυσμού είναι κάτω από 150 ε, λίρες την εβδομάδα. Πώς μπορείτε να εξηγήσετε λοιπόν στους ψηφοφόρους μου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ξοδεύει χρήματα των φορολογουμένων για πρόθεση, λέει, της Ευρωπαϊκής Ενότητας ή 411.000 ε, ευρώ για ένα κοινοτροφείο στην Ουγγαρία. Ενώ θα μπορούσατε να πληρώνετε και να θα είστε τους ψηφοφόρους μου. Θα μας υποσχεθείτε τουλάχιστον ότι θα πάψετε να ξοδεύετε τα χρήματά μας σε αυτά που εμείς στα West Midlands αποκαλούμε Yampi Schemes. Ευχαριστώ. Mm. Έχω αναλάβει αυτή την ευθύνη για τη σωστή απόδοση των ε, χρημάτων και αυτοί που είναι οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι θα πρέπει να καταβάλουν και τις μεγαλύτερες προσπάθειες και εσείς μετά την αποβιομηχάνηση ζήσατε μία μεγάλη κρίση. Ιδιαίτερα στη δική σας ε, περιφέρεια το ζήσατε αυτό. Και έπρεπε κανείς να αντιμετωπίσει της, ε, τη περιφέρεια αυτή η οποία βρέθηκε σε μία κατάσταση αποβιομηχάνησης. Ζήσατε μία μεγάλη παρακμή και νομίζω ότι με βάση τον, μεγάλο, τον νέο κανονισμό ορίζονται σαφή κριτήρια έτσι ώστε να μην γίνει κατασπατάληση πόρων. Διότι τα παραδείγματα που είπατε, ε, δηλαδή γήπεδα γκολφ, ε, κέντρα fitness, δεν δικαιολογούνται τη στιγμή που υπάρχουν περιφέρειες που δεν έχουν καν δημόσιες ε, τουαλέτες. Όλοι θέλουμε να πηγαίνουμε σε κέντρα fitness, αλλά δεν μπορούμε να τα χρηματοδοτούμε με κοινοτικά χρήματα, διότι υπάρχουν ε, μεγάλες ανάγκες για τους ανέργους και για αυτούς που χρειάζονται αυτά τα χρήματα. Και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτό τον τρόπο σκέψης Θέλουμε να καλύψουμε τις ανάγκες των πολιτών και τίποτα άλλο. Και αυτό περιλαμβάνει και πολλές ε, περιφέρειες του Ηνωμένου Βασιλείου. Ευχαριστώ. And the next question is from Κύριε Αουστερβίσιους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υποψηφία Επιτροπέ μετά από την οικονομική κρίση αντιμετωπίζουμε ακόμα τις επιπτώσεις της και ένας από τους χαμένους είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έμειναν έξω από τις ροές, οικονομικές ροές, από το ρευτό δηλαδή. Ατενίζοντας τώρα την Ευρώπη 2020 φοβούμε ότι ίσως να μιλούμε περισσότερο για την ικανότητα απορρόφησης παρά για επενδύσεις τι μέτρα θα λάβετε λοιπόν ως Επίτροπος για να περιορίσετε τη λεγόμενη απορροφητική ικανότητα αλλά με την αρνητική έννοια και να σπρώξετε τις επικοινωνικές επιχειρήσεις περισσότερο σε επενδύσεις. Δεύτερο, ποια νέα δημοσιονομικά εργαλεία θα προτείνετε να χρησιμοποιηθούν υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έτσι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε εύλογα ευρωπαϊκά κονδύλια. Θα βοηθήσουμε τις ΜΜΕ γιατί ε, οδηγούν στην ε, οικονομική ανάπτυξη. 70 δις ευρώ χορηγήθηκαν στις ΜΜΕ μεταξύ 7 και 14 Τώρα με τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές θα χορηγηθούν 140 δις ευρώ, δηλαδή θα διπλασιαστεί αυτό το ποσό. Βεβαίως ε, τα κράτη θα πρέπει και οι περιφέρειες θα πρέπει να απορροφήσουν αυτά τα ποσά και ελπίζω να μην βρεθούμε στη δυσχερή θέση του παρελθόντος όπου είχαμε ευφυή προγράμματα, καλά προγράμματα, τα οποία όμως δεν μπόρεσαν να απορροφήσουν αυτούς τους πόρους. Η απορρόφηση είναι πολύ σημαντική και θα ήθελα να ενθαρρύνω τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν με τις ΜΜΕ για να βρουν τον κατάλληλο τρόπο χρηματοδότησης γιατί έτσι θα βελτιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις της πολιτικής συνοχής. Thank you. And now I'll give a floor. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκέρικε. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ε, θα πρέπει να υπάρξουν ε, καλύτερες διοικητικές, διαχειριστικές ικανότητες. Ε, τα κριτήρια για την επιλεξιμότητα γίνονται όλα πιο σύνθετα. Τι θα κάνετε για να προωθήσετε την ε, απλοποίηση των προγραμμάτων και τη μείωση της γραφειοκρατίας τα, οι προποθέσει δεν είναι γνωστέ σε όλε τι περιφέρειε. Η Επιτροπή και οι χώρε μέλη και οι περιφέρειε χρειάζονται μεγαλύτερη ανταλλαγή εμπειριών. Τι θα κάνετε εσεί ω Επίτροπο για να ενισχύσετε αυτή την ανταλλαγή εμπειριών. Αν δεχθούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα χρηματοδοτήσει τη σύνδεση μεταξύ Δαλματίας ε, και Κροατίας, ε, τι θα κάνετε για να επιλύσετε το πρόβλημα αυτό στη μεθοριακή αυτή ε, περιοχή εάν ε, η Κροατία προσχωρήσει στη ζώνη Σέγγεν. Θα ήθελα να τονίσω ότι μειώθηκε η γραφειοκρατία από τους κανονισμούς που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι δεν απλοποιήθηκαν οι κανονισμοί. Αυτό που έχει σημασία είναι να βρούμε ακόμα 40 υπογραφές. Και αυτό εξαρτάται από κάθε χώρα. Αλλά θα πρέπει να εξεύρουμε αυτή την εξισορρόπηση μεταξύ απλούστευσης και ελέγχου. Δηλαδή ρύθμισης και νομιμότητας. Γιατί από τη μία πλευρά μιλάμε για απλουστεύσεις, αλλά υπάρχουν πολλές ε, φωνές για την... που μιλάνε για μεγαλύτερη αυστηρότητα από τους κανονισμούς. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τους δικαιούχους, αλλά να είμαστε πολύ προσεκτικοί με το πώς καταβάλλονται αυτά τα χρήματα. Δεν ελαχιστοποιώ τον παράγοντα αυστηρότητας η ευρωπαϊκή πολιτική προβάλλει ευκαιρίες, αλλά ξέρω ότι σε ορισμένες περιφέρειες δεν είναι, ε, δεν είναι ε, εύκολη η πρόσβαση. Ο κύριος Βανίστελ Ρόι έδωσε μεγάλο, μεγάλη μάχη και δεν ξέρω πώς ε, κάθε περιφέρεια θα μπορούσε να έχει υψηλή τεχνολογία. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Δηλαδή και οι λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες να δημιουργήσουν σημεία ε, που αποτελούν δέλεαρ. Δηλαδή η Ελλάδα με τη ΦΕΤΑ ε, ή άλλες χώρες με κάτι άλλο. Δεν πρέπει να είμαστε ένα Silicon Valley όλοι. Κάθε περιφέρεια έχει τις δικές της ε, δυνατότητες και θα πρέπει οι τοπικές αρχές να το δουν αυτό. Ακόμα και στις πιο φτωχές περιφέρειες υπάρχουν σχολεία, υπάρχουν πανεπιστήμια, υπάρχει δημόσια διοίκηση. Θα μπορέσουν να δούνε ποιο είναι το βασικό μας ατού. Η παλίνκα στην ε, Ουμπαρία, η τσουίκα στη Ρουμανία, η φέτα στην Ελλάδα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει σωστή πληροφόρηση για να ξέρουμε ποια είναι τα μπραντ μας. Στη Σεβίλια, στη Σεβίλη με συγχωρείτε, υπάρχει αυτή η πλατφόρμα καινοτομίας η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Η κάθε χώρα λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα ατού που διαθέτει. Thank you. Η πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση της κυρίας Βάνα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τελευταία ερώτηση, πράγματι, προστασία του κλίματος και η οικολογική αναδιάρθρωση της οικονομίας. Τον Ιούλιο που μας πέρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ανακοίνωση για την πράσινη οικονομία και για το υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό, ιδίως των αηφόρων ε, οικονομιών και των νέων πράσινων των εισαγωγικών θέσεων απασχόλησης. Και εκεί παίζουν ένα αρκετά σημαντικό ρόλο τα τα ταμεία. Θα είναι πολύτιμη η, συμβολή η συμβολή για την ε, πράσινη αναδιάρθρωση της οικονομίας. Αυτό πρέπει να γίνει και ταχύτερα μάλιστα για να εξασφαλιστεί το μέλλον. Ερώτηση, ποια συγκεκριμένα βήματα θα κάνετε για να εντάξετε την πράσινη οικονομία και να την ενισχύσετε μέσα στα πλαίσια των διαρθωτικών ταμείων. Ε, Ευχαριστώ. Στη νέα περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 η οικολογική αυτή διάσταση έχει μεγάλη σημασία. 38 δις εκατομμύρια θα αποδοθούν στην ενεργειακή αποδοτικότητα αλλά και στην οικολογική διάσταση της ενέργειας αυτό το αίτημα των πρασίνων θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα που σχετίζεται με την καθημερινή μας ζωή, τον τρόπο που ζούμε και πώς βελτιώνουμε το περιβάλλον όπου διαβιώνουμε εμείς και τα παιδιά μας. Θα δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Αλλά σας εγγυώμαι ότι δεν θα ξεχάσουμε αυτή την οικολογική διάσταση που είναι πολύ σημαντική. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη για τις ερωτήσεις και την υποψηφία επίτροπο για τις απαντήσεις. Πραγματικά ήταν ένα ε, δύσκολο, απαιτητικό πρωινό, αλλά επίσης πολύ χρήσιμο. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συμβολή σας. Πριν δώσω το λόγο στην υποψηφία επίτροπο για τις ε, καταληκτικές της ε, δηλώσεις, θα ήθελα να καλέσω τον ε, πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειών να κάνει μία δήλωση τριών λεπτών έτσι όπως ε, το συνηθίζουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης τα μέλη της, ε, Επιτροπ... της Περιφερειακής Επιτροπής και Κυρία Επίτροπε, βεβαίως για μας η πολιτική συνοχή είναι πρωτεύουσα σημασία γιατί ξέρετε ότι οι τοπικές αρχές τις οποίες εκπροσωπούμε είναι τελικά οι αποδέκτες του ε, περίπου 70% των διαφορετικών ταμείων. Η Επιτροπή Περιφερειών καλείται να διαδραματίσει το ρόλο ενός ενδιάμεσου μεταξύ ευρωπαϊκών και τοπικών αρχών. Και θα ήθελα εν συντομία να επιμείνω σε ορισμένα σημεία τα οποία είναι σημαντικά για μας. Η έκτη έκθεση για την ε, κοινωνική και εδαφική συνοχή προβλέπει ένα νέο εδαφικό όραμα στο πλαίσιο της αναθεωρημένης στρατηγικής Ευρώπη 2020 ε, και θα υπάρξει η λευκή βίβλος η οποία θα μας επιτρέψει να σημειώσουμε προόδους όσον αφορά την πολιτική συνοχής και μετά το 2020. Αναφέρθηκε εδώ το πρόβλημα των αστικών περιοχών και ελέγχθη ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει μια λευκή βίβλος, μια ολοκληρωμένη αστική ατζέντα ε, η οποία να επιτρέψει την ε, ολοκλήρωση της πολιτικής. Τα διαρθωτικά ταμεία 350 ε, δις θα συνεχίσουν να διατίθενται τι θα προτείνατε εσείς εκ μέρους της Επιτροπής ούτως ώστε να υποστηρίξετε μια μεγαλύτερη απορροφητικότητα των ε, πόρων από τις ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές γιατί ε, μπορούμε να προσεγγίσουμε το πρόβλημα αυτό μόνον εφόσον συνεργαστούμε και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με ΣΑΣΑ. Η Επιτροπή Περιφερειών ζήτησε να ενισχυθεί ο ρόλος των ε, περιφερειών και ε, προβλέπει βεβαίως το σύμφωνο σταθερότητας την ενίσχυση της ε, απασχόλησης στις πιο μειονεκτούσες περιοχές. Εμείς ε, πρόκειται να ορίσουμε και να ελοπίσουμε μαζί με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την, ε, μια στρατηγική αποκεντρωμένη επικοινωνία τη Ευρωπαϊκή Πολιτική, ούτω ώστε να εξηγήσουμε στου Ευρωπαίου πολίτε την προσθέμενη αξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ανοιχτές ε, ημέρες, οι οποίες διοργανώνουμε με την ε, Περιφερειακή Επιτροπή, συνιστούν μια μοναδική ευκαιρία για να γίνει κάτι τέτοιο. Για τις ε, γειτονικές, για τις χώρες, γιατί υπάρχουν σχέσεις με τη Νότια Μεσόγειο και την Ανατολική Ευρώπη εδώ η πολιτική αποκέντρωση οδηγήσε στην ενίσχυση των δεσμών με τις ε, τοπικές αρχές υπέρ της αύξησης και της δημιουργίας των θέσεων απασχόλησης. Κυρία υποψηφία Επίτροπε, ε, ε, ε, χαίρομαι πάρα πολύ που εξαγγείλετε την ε, δέσμευσή σας να γίνετε μια πρέσβυρα υπέρ της, ε, των αστικών περιοχών και των περιφερειών. για την Επιτροπή Περιφερειών, εκ μέρους της Επιτροπής Περιφερειών θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που προτίθεστε να εφαρμόσετε μια αρχή την οποία και εμείς στηρίζουμε την αρχή της ε, διακυβέρνησης. Παρακαλώ. Η κυρία Κρέτσου, υποψήφια επίτροπος. Ας προβεί στην σύντομη καταληκτική της ε, δήλωση που να μην υπερβεί τα πέντε λεπτά. Θα είμαι και συντομότερη των πέντε λεπτών, κυρία Πρόεδρε. Γνωρίζω ότι μακρηγόρησα τις απαντήσεις μου. Μιλήσαμε τρεις ώρες τώρα σε τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση για την πολιτική συνοχή. Έχω κάποιες σκέψεις ωστόσο που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Ήταν συναισθηματικά φορτισμένη η περίοδος αυτή των ε, τριών ωρών, αλλά ήμουν και οκτώ χρόνια εδώ. Άρχισα ένα χρόνο πριν να ενταχθεί η Ρουμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως παρατηρήτρια. Και θυμούμε, σαν ήταν χθε, την πρώτη μέρα που εισήλθα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα συναισθήματα που με διακατήχαν όταν έγινα για πρώτη φορά ευρω, ευρωβουλευτής. Θα ήθελα να σας πω ότι θα ήταν πολύ δυσκολότερο για μένα να είμαι σήμερα ενώπιόν σας χωρίς την τεράστια εμπειρία που απέκτησα στη διάρκεια των 8 αυτών ετών ως ευρωβουλευτής. Ορισμένοι εξημών με γνωρίζετε. Όπως ήμουν θα παραμείνω. Θα ήθελα να διατηρήσω και τις ίδιες σχέσεις μαζί σας που είχαμε πάντοτε. Γνωρίζω σε ό,τι αφορά την δική σας επιτροπή τις θετικές εμπειρίες που είχαμε. Πάντοτε θα θέλω να ανταλλάξω απόψεις μαζί σας και να λαμβάνουμε από κοινού αποφάσεις. Γιατί πρόκειται για πολύ σημαντικό τομέα και είναι πολύ σημαντικό να εργαστούμε μαζί προς το συμφέρον των πολιτών και της Ευρώπης γενικότερα. Σας βεβαιώνω ότι εάν τελικώς διοριστώ επίτροπος θα αγωνιστώ υπέρ των ίδιων αξιών υπέρ των οποίων εργαστήκαμε και μαζί ως Ευρωβουλευτές όλα αυτά τα χρόνια. Αξιοπρέπεια, ή μεταχείριση για όλες τις χώρες μέλη. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ και πάλι και πάντοτε θα προσέρχομαι ενώπιον σας με ιδιαίτερη χαρά κάθε φορά δηλαδή που θα θέλετε ε, να με δείτε και βεβαίω όταν θα έχετε κρίνει πρώτα περί της μοίρας μου. Ευχαριστώ. Thank you. Thank Η Πρόεδρος Μιχαήλοβα, ευχαριστώ και εσάς κυρία Κρέτσου και όλα τα μέλη. Η συνάντηση για την αξιολόγηση των συντονιστών που θα γίνει σήμερα το απόγευμα και κλεισμένων των θυρών από τη μία μέχρι τις δύο απογευματινές ώρες στο 4Β001, αίθουσα 4Β001 και τώρα εδώ λίγη συνεδρίαση.